Uh, good morning, ladies Νομίζω ήμουν γενναιόδωρος, επιτρέποντας χρόνο για να καθίσουν για τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς αυτή τη βδομάδα, όπου έχουμε δύο ιδιαίτερα θέματα. Την παρουσίαση του κυρίου Σουβάμπ, που αδειμονούμε να ακούσουμε, να δούμε αυτή την έκθεση για την οδηγία περί δικαιωμάτων των καταναλωτών και που αναμένουν και οθόνες τις ιδέες να υποβληθούν. Και θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα για τα όσα έγιναν στη συνάντηση συντονιστών χθε και κάποιες αυσκυριότερες αποφάσεις. Φυσικά όλα τα μέλη της Επιτροπής θα πάρουν ένα σημείωμα για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές μέσα στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, ως ήθιστε. Να σας πω ότι δύο γνωμοδοτήσεις προς άλλες συναυλευτικές επιτροπές θα συντάξουμε. Έχουμε μια δική μας έκθεση διασπορτοβουλίας, Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, νομίζω. Α, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Συγγνώμη, συντάσσει μια έκθεση για το πρόγραμμα δράσης όσον αφορά το πρόγραμμα Στοχόλμης. Και ένα μέλος της, ε, των σοσιαλιστών θα συντάξει αυτή τη γνωμοδότηση. Μια δεύτερη γνωμοδότηση όσον αφορά την μείωση των ανισοτήτων στην υγεία σε σχέση με την ε, ομάδα ECR θα λάβει αυτή, αυτή τη γνωμοδότηση. Οι συντονιστές λοιπόν θα διορίσουν ένα συντάκτη σχετικά σύντομα. Οι συντονιστές συμφώνησαν επίσης ε, ότι θα ζητηθεί μια νέα έκθεση ιδιαίτερη για την παρακολούθηση του τομέα λιανικού εμπορίου. Παράλληλα με το έργο που ε, γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής και αναμένουμε να έχουμε και μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτό. Βρίσκεται λοιπόν μπροστά η Επιτροπή από, στο παιχνίδι σε σχέση με την τοποθέτηση επί πολιτικών θεμάτων. Οι συντονιστές συμφώνησαν για ένα αίτημα Μόζαρ για την ε, οδηγία περί ασφάλειας και όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και για ένα workshop σεμινάριο 28-29 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί. Έχει συμφωνηθεί η χρονική στιγμή. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον κύριο αυτό και θέλω πάλι να αναφέρω ότι έχουμε εδώ πάλι μια έκθεση όπου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζει τα πολιτικά θέματα γύρω από τα θέματα αυτής της οδηγίας και αναμένοντας την πρόταση το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να γνωρίζετε ίσως ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες να δοθούν κάποιες ε, παρατηρήσεις, ε, σχόλια, παρεμβάσεις ε, ήδη εκ προημίου, πράγμα το οποίο είναι καλοδεχούμενο όσον αφορά το νομοθετικό έργο. Και τέλος να σας αναφέρω ότι συνεχίζουμε με τη διοργάνωση ενός φόρουμ για την ενιαία εσωτερική αγορά. Μια από τις σημαντικές συστάσεις ε, των εκθέσεων των και Γκρέκ για τα θέματα εσωτερικής ε, αγοράς ε, και τα σχέδια αυτά είναι υπό αίρεση έγκρισης από πλευράς Προέδρου Κοινοβουλίου σε 9 Νοεμβρίου το απόγευμα. Σε συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία θα διοργανωθεί και ελπίζουμε ότι θα γίνει στην αίθουσα Αλομέλειας στο ημικύκλιο και ότι ενθουσιώδης θα είναι η συμμετοχή και θα συναθριστούν πολλοί πληθώρα ευρωβουλευτών. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Και έτσι λοιπόν με αυτά πρωτού καλέσω τον κύριο Σβάμπ να μας παρουσιάσει την έκθεσή του στο πρώτο σημείο. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Νταϊάννα Γουόλης, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου ιδιαίτερα ενεργό μέλος ε, της ε, ε, αντίστοιχης επιτροπής και ηγέτης αδιαμφισβήτητα για το κοινό πλαίσιο αναφοράς θα έλεγα. Με ιδιαίτερη χαρά σας βλέπουμε εδώ κυρία Γουόλης και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεισφέρετε θετικά στη συζήτηση και από πλευρά σας. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων. <clears throat> Η οδηγία περί δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι χωρίς αμφιβολία το πιο σημαντικό νομοθετικό τμήμα του έργου της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής επί μακρόχρονικό διάστημα και είχαμε και σεμινάρια και αναλύσεις και τώρα περνάμε στο σημείο όπου ο εισηγητής μας κύριος Ανδρέας Σβάμπ θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία αποκαλύπτοντας τις προτάσεις του. Με τα επτά πέπλα της Σαλόμης θα αποκαλυφθούν τώρα όλα τα στοιχεία και θα μας εξηγήσει την αλληλουχία των γεγονότων που πρέπει να καλυφθούν. Έχετε τον λόγο κύριε Σβάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και για αυτές τις, ε, αυτούς τους επένους που μου δώσατε ενώ ξεκινά μόλις η εργασία. Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και τη γραμματεία να τους ευχαριστήσω διότι η παρουσίαση, η παρουσίαση λέω του κειμένου που σήμερα είναι στη διάθεσή μας ήταν δυνατό να γίνει με αυτόν τον τρόπο έχοντας μια σύνοψη κειμένου, μια περιεκτική έκδοση του κειμένου. Ήταν εφικτό αυτό για τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες για να δοθεί μια σύνοψη στους συναδέλφους τι αλλάζει τώρα και πόσα και πού απορρέουν αυτές οι, οι τροποποίησεις. Δεύτερον, ευχαριστώ τη Γραμματεία και τους μεταφραστές για μια σημαντική επίδοση. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι το γαλλικό κείμενο το οποίο διάβασα έχει κάποια σημαντικά σφάλματα παρόλα αυτά. Το 14 μεταφράστηκε με 15 και δεν μπορώ δυστυχώς να διασφαλίσω ότι όλα είναι σωστά. Πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα της, ε, των γλωσσικών των μεταφράσεων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, την κυρία Βερνιό, τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν για το πράσινο βιβλίο, την κυρία Μακάρθη και πολλούς πολλούς άλλους συναδέλφους που σημαντικές ε, παρεμβάσεις έκαναν από πλευρά του. Ξεκινώντας θα ήθελα σύντομα να υπενθυμίσω ποιες είναι οι βασικές αρχές που μας απασχόλησαν Θέλουμε το επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να αναβαθμιστεί θέλαμε να υπάρξει εξαπλούστευση και ενιαίο πλαίσιο των κανόνων για την προστασία καταναλωτών. Γιατί μόνο η διαφάνεια για τα δικαιώματα των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει σε γνώση, σε αντικειμενική γνώση. Και μόνο όποιο γνωρίζει τα δικαιώματα του μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα αυτά και να επιβάλλει το σεβασμό του. Ταυτόχρονα και η υποστήριξη που, τις οποίες τύχαμε από πλευρά τη Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή, ότι δηλαδή οι καταναλωτέ στην ενιαία εσωτερική αγορά μέσω ενό μεγαλύτερου, ακόμα μεγαλύτερου φάσματος θα πρέπει να προστατεύονται. Και όταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνουν τέτοιου είδους διασυνοριακές προσφορές για συναλλαγές, ώστε η πολιτισμική και η οικονομική πολυμορφία της Ευρώπης να διασφαλιστεί. Για την νομική ασφάλεια, αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο όταν έχουν 20.000 ευρώ ετήσια τα οποία επενδύονται στη συνεθνική αγορά και 400.000 ευρώ θα πρέπει να ε, είναι ο τζίρος προτού τολμήσουν να περάσουν σε διασυνοριακές συναλλαγές αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συζήτηση στην Επιτροπή μας έδειξε ότι διακομματικά συμφωνούμε. Η πρόταση αυτή όπως υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεν βρίσκει τη συνένεσή μας και γι' αυτό πονήσαμε μια νέα αναθεώρηση αυτής της πρότασης εκ Μια πλήρη αναθεώρηση κάναμε έδωσα την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πρόταση που νομίζω σε πολλά σημεία αντανακλά αυτά τα οποία στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή συνενετικά ζητήσαμε όλοι. Και γι' αυτό θα ήθελα συγκεκριμένα να περάσω τώρα σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία σας υποβάλλω και εξηγώ για κατανόηση από πλευρά σας. Αντίθετα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται στις, στην, στην 8η ε, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 8 αυτές οδηγίες και τέσσερις από αυτές που πρέπει πλήρως να αντικατασταθούν, η δική μου πρόταση τι κάνει αναφέρεται σε, μια ε, ρύθμιση ομπρέλας ε, που θα ρυθμίζει όλα αυτά τα θέματα. Τις τέσσερις εκείνες ε, που επιλέγει από τις οδηγίες αυτές όπου στοχοθετημένα συμφωνούμε και συνενούμε για μια απλούστευση στοχοθετημένη όμως Όλα τα άλλα θέματα παραμένουν στις ε, οδηγίες ε, ως βάση και έτσι μέσα στο πλαίσιο του ελάχιστου εναρμονισμού αυτή η συστέγαση, α το πω έτσι, σφαιρική ρύθμιση αφήνει τη δυνατότητα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή στι διαβουλεύσει να έχουμε μια ελαστικότητα. Τι θα εντάσσεται δηλαδή, τι δεν θα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να μην τροχοπεδηθεί η πρόταση όταν έχουμε κάποια δισκαμψία. Να έχουμε μια ελαστικότητα, τι θα ε, ρυθμιστεί συνολικά και τι όχι. Ταυτόχρονα όμως να, είχα, να έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο των ε, θεμελιωδών οδηγιών να κάνουμε κάποιες αλλαγές ε, όσον αφορά τον ελάχιστο εναρμονισμό. Ταυτόχρονα μια τεχνική ρυθμίσεων για το μέλλον που αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα απλούστευσης για το μέλλον. Διότι αυτή η σφαιρική συνολική ρύθμιση στο μέλλον νέα στοιχεία για την εξαπλούστευση επιτρέπει να εισαχθούν και να ε, λειτουργήσουν. Ο στόχος ή το στόχο μας το περιέγραψα ως εξής. Πρόκειται ουσιαστικά και για τα δύο. Βελτίωση της ε, ε, προσφοράς ε, διασυνοριακά, βελτίωση της αποτελεσματικότητας, υπήρξε συνένεση σε σχέση με αυτά τα θέματα και χθε με την έκθεση Παύλο Άριας. Με τον, την απλούστευση έχουμε την εξή διαχωριστική γραμμή. Η κυρία Πίτροπο Ρέντινγκ, την οποία και για την ελαστικότητά τη, μεγάλη ελαστικότητα, την ευχαριστώ σε αυτή την πρόταση, ή χρησιμοποίησε την έννοια face to face ω διαχωριστική γραμμή, ενώπιο ενωπίο. Θα έλεγα ότι με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής σε κάποιο, κατά κάποιο τρόπο ε, ισοπεδώνεται πολλές φορές ε, και για θέματα τα οποία έχουν σημασία. Αυτή την κατάσταση πρέπει να τη ρυθμίσουμε όμως εμείς. Ταυτόχρονα πρέπει να δεχθούμε όμως ότι υπάρχει μια ευρεία πλειοψηφία κατά της ρύθμισης όλων αυτών των συμβάσεων ή συμβατικών στοιχείων. Γι' αυτό και στο πράσινο και στο κόκκινο κουτί θα δείτε ποιες ρυθμίσεις υπάρχουν όσον αφορά τον στόχο του πλήρους εναρμονισμού, δηλαδή όλες οι τηλεσυμβάσεις, distance contracts, δηλαδή δεν έχουμε διαχωριστική γραμμή το face-to-face ενώπιος ενώπιο, αλλά off-premises και on-premises. Δηλαδή σε κλειστό ή σε ανοιχτό τηλε ή εκ του σύνεγγυς ε, τέτοιες επαφές. Και έχουμε και το 80% συνολικά αυτών των συμβάσεων που θα παραμείνουν σε εθνικό ε, νομικό πλαίσιο. Και έχουμε και στο 4β περαιτέρω συμβάσεις που εξαιρούνται από τον πλήρη εναρμονισμό. Για παράδειγμα, κοινωνικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή θέματα μεταφοράς, για παράδειγμα επιχειρήσεις ταξί και άλλα συναφή υπό το άρθρο 4β μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά. Στο επόμενο τώρα χαρτί μπορεί κανείς να δει τη δομή της δικής μου πρότασης σήμερα πώς έχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν πέντε κεφάλαια είχε προτείνει εγώ διατήρησα σε μεγάλο βαθμό αυτή τη δομή. Το κεφάλαιο 1 κάπως το επεξέτεινα. Θα ήθελα να σας προτείνω το, τα κεφάλαια 2 και 3 με αυτή την καλύτερα στοχοθετημένη ε, πρόταση να τα συγχωνεύσουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη ρύθμιση. Επειδή το off-premises και distance selling contracts θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης. Και στο κεφάλαιο 5, μεγάλες αλλαγές μετά από τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή, μεγάλες αλλαγές έγιναν. Στο κεφάλαιο 6 προτείνω τυπικά και επίσημα κάποιες προτάσεις που τις διαδικασίες ε, ε, σε σχέση με αυτή την πρόταση που δεν ήταν πολύ ευτυχής, πολύ καλές μπορούν να βελτιωθούν. Και όσον αφορά το κεφάλαιο για το πεδίο εφαρμογής και ορισμούς, με την ένταξη κανόνων, και η κυρία Γόλης είναι παρούσα, κανόνων για το κοινό πλαίσιο αναφοράς, δημιουργούμε μια βελτιωμένη κίνηση για την ε, προσπελασιμότητα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και είμαστε υπέρ ενός νέου άρθρου 2α, μια καλύτερη συνεκτικότητα με άλλα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα καταναλωτών στην ενιαία εσωτερική αγορά. Έτσι δημιουργούμε έναν ενιαίο ορισμό των ε, ε, τηλεπολίσεων, για παράδειγμα, της τηλεεμπορίας. Έχουμε επίσης και την παροχή, των, την παροχή υπηρεσιών που αλλού ρυθμίζονται στο κεφάλαιο 2 που είναι πράσινο επειδή βασίζεται στην αρχή του πλήρους εναρμονισμού και έτσι τις οδηγίες που έχουμε σε βάση και που προηγούμενα αναφέραμε distance selling και doorstep selling τις αντικαθιστούν πλήρως οι προτάσεις εδώ Προβλέπεται λοιπόν εδώ μέσω της συγχώνευσης ε, του πεδίου εφαρμογής ε, χρειαζόμαστε λιγότερο εύρος, με συγχωρείτε. Και έτσι καταφέρνουμε μέσα σε περιεκτικό, με περιεκτικότερο τρόπο να είμαστε πιο ευανάγνωστοι. Έχουμε το κόκκινο και πράσινο στη συνέχεια. Στο, ο κόκκινος τομέας είναι ο τομέας της ελάχιστης ε, εναρμόνισης. Ενώ κάποια σημεία τα οποία αναφέρονται εδώ τα θέτουμε σε ένα ξεχωριστό, σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο για ε, ξεχωριστή στοχοθέτηση. Στο κεφάλι 4 δεν νομίζω ότι υποβάλλω, θα υποβάλλεται μια πρόταση όσον αφορά τα τέλη Ιουλίου, Ιουνίου με συγχωρείτε, για την απλούστευση των δικαιωμάτων ε, παροχής, αλλά τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στο επίπεδο του ελάχιστου εναρμονισμού. Θα ήθελα κυρίω εδώ να σα δώσω μια σύνοψη συνολικά για αυτή την οδηγία, για να μπορέσετε να εξοικειωθείτε σε ποιου τομεί, ε, με ποιο στοχοθετημένο τρόπο ε, βασίζονται σε απλούστευση οι προτάσει και σε ποιου τομεί βασίζονται στον ελάχιστο εναρμονισμό. Δηλαδή το νέο κεφάλαιο 2, με άλλα λόγια θα είναι πράσινο και τα κεφάλαια 4 και 5 παραμένουν κόκκινα-πράσινα και κόκκινα και πράσινα. Για τις λεπτομέρειες ιστερότερα, ε, μεταγενέστερα θα συζητήσουμε. Αυτό προτείνω για τα κεφα... τις ε, λεπτομέρειες των κεφαλαίων 2 και 1 μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Για τα κεφάλαια 2 και 3 θα ήθελα κάποιες άλλες λεπτομέρειες να αναφέρω επιπρόσθετα. Το νέο άρθρο 5 δεν ξέρω τώρα αν είναι εδώ το γράφημα διαθέσιμο μια και δεν αλλάζει. Α, είναι, άλλαξε, είναι εδώ, εντάξει το έχουμε. Ε, υπέβαλα μια πρόταση για τις απαιτήσει για την πληροφόρηση σε σχέση με τις συμβάσεις που θα συντάσσονται. Είναι σημαντικό ότι ζήσαμε μια σειρά περιπτώσεων όπου οι εμπορευόμενοι, οι επιτιδευματίες πολλά στοιχεία δεν ε, τα διαβίβαζαν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που μετά από την κράτηση δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό ή κάποιο, κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υπάρχει επαφή. Εδώ θα ήθελα να προτείνω να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρησης να είναι δεσμευτική και έτσι να χρειάζεται ο, παρέχουν την υπηρεσία δεσμευτικά να αναγκάζεται αυτά τα στοιχεία να τα διασφαλίζει. Στην ε, ε, υποχρέωση πληροφόρησης υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν. Με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους που ενδιαφέρονται συζήτησα υπάρχει μια βεβαιότητα αν στον τομέα των υποχρεώσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης μπορεί να υπάρξει στοχοθέτηση, διότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν δυσκολίες ο συνάδελφος βοηθός που προέρχεται από την Αυστρία. Στην Αυστρία υπάρχει ένα νομοθέτημα που προβλέπει ότι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα τατουάζ, αυτό άκουσα τουλάχιστον, όσοι θέλουν να κάνουν ένα τατουάζ, ε, έχουν πρόσθετη υποχρέωση ε, πληροφόρησης. Εγώ δεν έχω ε, κάτι τέτοιο υπόψη να καταστήσω υποχρεωτικό να καταργηθεί μια τέτοια ρύθμιση διότι αυτές οι ε, ρυθμίσεις βασίζονται στην αποφυγή κινδύνων όσο αφορά την υγεία. Και εδώ έχουμε και τον τομέα της δημόσιας τάξης, ε, την υγεία και το περιβάλλον ως στοιχεία τα οποία ρυθμίζονται από τα κράτη-μέλη και εξαιρούνται. Αφήνουμε όμως τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ισχύουν τέτοιοι κανόνες. Στη Γαλλία υπάρχει η συζήτηση αν ε, εδώ δεν συγκρούονται κάποιες διατάξεις και εδώ πάλι ε, ισχύει η αρχή ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν αυτές τις διατάξεις. Δεύτερον, ήταν σημαντικό αίτημα της Οικονομικής Επιτροπής που χτες ε, υπέβαλε τη δική της γνωμοδότηση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στο χρηματοοικονομικό τομέα προσπαθούν να γεμίσουν, να καλύψουν κάποια κενά. Και εδώ υπάρχει μια μικρή σειρά ασφαλίσεων ή παροχών όσον αφορά συμβάσεις ε, στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι αυτές οι ε, συμβάσεις που ε, συνάπτονται εκτός δεδομένων πλαισίων και δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ όμως η Οικονομική Επιτροπή συνενετικά ζήτησε η, η δυνατότητα εφαρμογής να προβλέπεται στις διατάξεις από πλευράς μας. Τρίτον, θα ήθελα ενιαία πρότυπα ερωτηματολογίων ή ε, εγγράφων που θα συμπληρώνονται να ισχύουν. Ευρωπαϊκά, πανευρωπαϊκά να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργείται ένας ευνοϊκός όρος να συμπληρώνονται αυτά τα ενιαία ε, έγγραφα, έντυπα και να μην επιβαρύνονται ιδιαίτερα. Επίσης ε, καθορίστηκε ότι η δυνατότητα ανάκλησης θα προβλέπει περίοδο 14 ε, ημερολογιακών ημερών. Είναι σημαντικό αυτό, διότι επεκτείνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών πανευρωπαϊκά. Αν ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί σωστά για τα δικαιώματά του, χρειάζεται κάποιο στοιχείο κύρωσης, κάποια ποινή ε, για το ότι δεν συνέβη αυτό. Γι' αυτό σας προτείνω σε τέτοιες περιπτώσεις που στα κράτη-μέλη με πολύ διαφορετικό τρόπο και έχουμε κάποιες ε, εβδομάδες ε, περίοδου διορίας να έχουμε ένα έτος ένα έτος ώστε να υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης από πλευράς ε, ενός ε, καταναλωτή όταν θα έχει αποδειχθεί η μη ε, τήρηση αυτών των στοιχείων. Επιπλέον προσπάθησα πρακτικές δυνατότητες να δημιουργήσω τοπικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χειροτεχνία τους χειρόνακτες, σε μια κατάσταση, για παράδειγμα, όταν κάποιος καλείται να παράσχει μια υπηρεσία, αυτού του είδους οι υπηρεσίες που με πρακτικό τρόπο πρέπει να παρέχονται, να μπορούν με την μεγαλύτερη ελαστικότητα να αντιμετωπίζονται και οι τοπικές υπηρεσίες χειρονακτών να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή επιβαρύνσεις, να εξαιρούνται από γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Σε κάποιου τομεί αυτό συνδέεται με κάποιε δυσκολίε, διότι προέβλεψα οι καταναλωτέ να έχουν ένα, μια δυνατότητα ανάκληση ε, όταν ε, παρέχονται υπηρεσίε από ένα οργανωμένο σύστημα. Πρέπει να μπορεί κανεί να, να διασφαλίσει ότι ε, το βάρος της απόδειξης δεν θα το έχει ο καταναλωτής, αλλά παρέχον την υπηρεσία. Και έτσι θα πρέπει εδώ να δούμε συνολικά το τι θα ισχύει σε σχέση με αυτές τις ε, υπηρεσίες. Τελευταίο σημείο, επέκταση σε άλλους τομείς. Αφήσαμε να ε, ισχύει το ότι για όλες τις αγορές αγαθών για οποιαδήποτε αγαθά θα ισχύουν αυτές οι διατάξεις ε, από ε, το κόστος της επιστροφής θα πρέπει από τον ε, εμπορευόμενο να καλύπτεται αν πρόκειται για τιμή άνω των 50 ευρώ σε σχέση με το αγαθό ή το προϊόν. Συμφωνούμε ότι όσοι πολλούν κάτι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης όσον αφορά τους πελάτες. Ακριβώς οι κρατήσεις όσον αφορά τα πτήσεις ε, θα πρέπει σε σχέση με την ε, διασφάλιση της ενημέρωσης των στοιχείων να διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Να μην είναι να μην είναι τυχαία, αλλά όλα, όλες οι πρόσθετες δαπάνες ε, και το κόστος να αποτελούν αντικείμενο ενημέρωσης σε σχέση με τον πελάτη από τον πάροχο. Θα καταλήξουμε σε αυτό και ολοκληρώνοντας σε σχέση με τις διαφημίσεις τις τηλεφωνικές. Οι τηλεφωνικές διαφημίσεις δεν απαγορεύονται με αυτήν την οδηγία. Υπάρχει ε, στην Γερμανία ένα ε, πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές διαφημίσεις. Αν όμως επιτρέπονται τέτοιου είδους διαφημίσεις από τα κράτη-μέλη ή παραμένουν σε ένα επίπεδο ε, που επιτρέπουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, τότε θα πρέπει στο αντίστοιχο άρθρο να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα και πάλι θα έχει το βάρος της απόδειξης ο πάροχος ότι έχουν, έχει δώσει τα σωστά πληροφοριακά στοιχεία στον πελάτη. Πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες κυρίες και κύριοι και γι' αυτό ενδιαφέρομαι άμεσα να ακούσω τις δικές σας απόψεις σε αυτή την πρόταση. Ξέρω ότι πολλά σε αυτή την πρόταση μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περαιτέρω και χαίρομαι ότι για τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό από κοινού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, well, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. που μας παρουσίασες τις πολύ σημαντικές αλλαγές που προτείνεις και νομίζω πως είναι καλή ιδέα Είναι καλή ιδέα να δούμε τις διαδικασίες και όλες τις ε, λεπτομέρειες. Ε, βέβαια δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σε σχέση με το πρόγραμμά μας θα εξετάσουμε τα 4 και το 5 στις 24 Ιουνίου και βέβαια θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα μας πούν ε, οι συνάδελφοι σήμερα και τα 6 και 7 στις 12 Ιουλίου. Και θα έχουμε προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 9 Σεπτεμβρίου και το Σεπτέμβριο για να δουλέψουμε πάνω στις τροπολογίες και στην Επιτροπή μας θα το δουλέψουμε ξανά στις 26 Οκτωβρίου. Έχουμε δώσει αρκετό χρόνο για να σκεφτούμε τα διάφορα στοιχεία γιατί είναι πολύ περίπλοκη αυτή η οδηγία. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους Κεώδης και στους υπόλοιπους ε, συναδέλφους να καλωσορίσω και το Συμβούλιο και την Επιτροπή εδώ. Δεν είμαι βέβαιος για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν. Α, ο κύριος Πρόγκ. Επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Κάλλος Κρέσπο από το Συμβούλιο που παρακολουθεί στενά τις εργασίες μας και ευχαρίστω να του δώσω και το λόγο αργότερα για να μας πει δύο λόγια για την πρόοδο ε, στο Συμβούλιο. Έχουμε και τον κύριο Πατάια από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την οποία, τον οποίο καλωσορίζω για να μας πει δύο λόγια για τη δική τους ε, ε, θέση. Τώρα, στις 10 έχουμε ψηφοφορία. Ίσως θα πρέπει να διακόψουμε τη συζήτηση, να κάνουμε τις ψηφοφορίες. και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μετά την ψηφοφορία. Ξέρω πως μπορεί να σας ε, δυσκολέψει κάπως, αλλά συνήθως ψηφίζουμε στις 10. Α κάνουμε λοιπόν ένα γύρο των σκιωδών εισηγητών. Καταρχήν η κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριος Ρόσφορ, η κυρία Τούνεν και εγώ θα αντικαταστήσω τον κύριο Μπίλαντ που είναι ο δικό μα σκιώδη, ο κύριο Τενταφυλίδης και ο κύριο Σαλβίνη, δεν τον βλέπω, είναι εδώ. Και μετά έχουμε την κυρία Βένιου και την κυρία Βόλης ε, ως ομιλητές. Και ίσως ε, χρειαστεί να σας ζωρίσω λίγο με το χρόνο, να σας πιέσω, εξαρτάται από το πόσο χρόνο θα έχουμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την ε, κυρία Γκέμπχαρτ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σουβάμπ για την παρουσίαση Τη δική σας πρόταση. Πρέπει να πω καμιά φορά με εκπλήσετε κύριε Σουβάμπ. Δεν ήξερα ότι είσαστε παδό ε, της πράσινης κόκκινης ε, κοινοβουλευτική συμμαχία. Γιατί όχι, συμπαθέστατη αυτή η προσέγγιση. Θα έλεγα λοιπόν ότι εσείς με αυτή την πρόταση που μας θέτετε επί τραπέζης, υπάρχει ανάγκη μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά. Το ξαναλέω για να το υπενθυμίσω αυτό, ότι εμεί ως κοινοβουλευτική ομάδα πάντα λέγαμε ότι το χαιρετίζουμε πολύ μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση του δικαιακού πλαισίου να μπορέσει να λειτουργήσει. Απλούστευση που θα διασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση και πιο εύκολη πρόσβαση και για τους επιχειρηματίες και για τους καταναλωτές στην ίδια την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενιαία εσωτερική αγορά, ώστε να μπορέσουν να διασφαλιστούν αυτά τα δύο. Ωστόσο όμως πάντα λέγαμε και Νομίζω εδώ συμφωνούμε μεταξύ μας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτρέψει να οδηγηθούμε το δικαίωμα για την προστασία των καταναλωτών θα υποβαθμιστεί και δυστυχώς συνέβη αυτό με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώς με αυτή την προσέγγιση του πλήρους εναρμονισμού από πλευράς της. Και γι' αυτό χαιρετίζω ακριβώς το ότι η κυρία Ρέντινγκ με σαφέστατο τρόπο είπε και χθε για παράδειγμα και όλα στο φόρουμ για την προστασία των καταναλωτών. Για άλλη μια φορά κατέστησε σαφέ η κυρία Ρέντινγκ ότι είναι υπέρ αυτός ο πλήρη εναρμονισμός να μην λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο όπως προβλέπεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να έχουμε μια ελαστική αντιμετώπιση και ότι είναι πρόθυμοι να συζητήσουμε, να συζητηθούν αυτά τα θέματα όλα και ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο για μια τέτοια πρόταση πλήρους εναρμοσμού δεν υπάρχει πλειοψηφία, διότι συνδέεται με μείωση, με υποβάθμιση της προστασίας των καταναλωτών. Είναι λοιπόν μια καλή προσέγγιση αυτή τώρα. Έχετε τώρα εσείς υποβάλει μια πρόταση επί τραπέζης που μόλις χθε την πρωτοείδα. Την πήρα στα χέρια μου χθε για πρώτη φορά. Δεν είχα φυσικά χρόνο μέχρι σήμερα το πρωί να τη μελετήσω σε βάθος. Εντάξει. Και Ήδη το είχατε προαναγγείλει σε συζητήσεις που είχαμε πιο πριν ότι κάτι τελείως καινούριο και νέο θα υποβάλλατε ως πρόταση σε σχέση όχι δηλαδή με μια σφαιρική πρόταση πλήρους εναρμονισμού αλλά μια προσέγγιση ελαστική με δυνατότητα αντιμετώπιση με ελαστικό τρόπο αυτών των τεσσάρων οδηγιών. Το πρόβλημα το οποίο τώρα βλέπω για να υπάρχει πλήρη κατανόηση αυτή τη πρότασή σα είναι ότι η πρότασή σα σας σταματούν οι προτάσει σα στο άρθρο 20. Οι άλλοι τομεί δεν είναι ακόμα στη διάθεσή μα. και είναι φυσικά πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς τι θα γίνει συνολικά με μια τέτοια προσέγγιση για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Θα υπάρχει μια ρύθμιση. Μπορεί να ακολουθηθεί μια τέτοια προσέγγιση ή θα έχουμε προβλήματα. Μια και τουλάχιστον στα πρώτα 20 άρθρα τα οποία αναφέρεται υπάρχουν αναφορές σε άρθρα που ακολουθούν μετά το άρθρο 20 και έτσι δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και να κατανοήσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της δικής σας πρότασης σε λεπτομέρειες. Είπατε επίσης ότι είναι σημαντικό για σας ότι η προστασία των καταναλωτών δεν πρέπει να υποβαθμιστεί. Εντάξει, έχω όμως την εντύπωση και ίσως είναι λανθασμένη η εντύπωσή μου αλλά αυτό πρέπει να το ελέγξουμε ότι σε ένα ή άλλο σημείο δεν δικαιώνεται αυτή την άποψή σας να μην υποβαθμιστεί η προστασία των καταναλωτών. Σε κάποιες προτάσεις, για παράδειγμα στα άρθρα 10 και 11 Ακολουθείτε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν ήδη χειρότερες σε σχέση με το σημερινό ενισχύει δίκαιο. Πάλι υποβαθμίζονται λοιπόν εδώ σχετικά κάποια θέματα και αν όλα αυτά επαληθεθούν στον έλεγχο, <laughs> στην εξέταση, εμείς ως κοινοβευτική ομάδα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά όπως λέω σε βάθος. Δεν είχα τη δυνατότητα μέχρι τώρα να τα εξετάσω πλήρως. Τώρα, ακριβώς από πλευράς του Προέδρου, Αναφέρθηκε και η χρονική ε, προθεσμία ή συνιστόσα. Αν βλέπουμε σωστά τα πράγματα, το τελευταίο τμήμα του σχεδίου έκθεσής σας στις 12 Ιουλίου θα το έχουμε μπροστά μας. Έτσι. Πολύ στερότερα δηλαδή. Ή για πρώτη φορά τότε θα το συζητήσουμε, πώς να το πω. Και για τα κεφάλαια 6 και 7, έτσι. Ε, αυτό έγινε κατανοητό. Ο κύριος Πρόεδρος όμως είπε ότι κατά τα τέλη Ιουνίου τα κεφάλαια 4 και 5 και μετά 6 και 7 τον Ιούλιο που θα ακολουθήσουν θα συζητηθούν. Αυτό δεν είπατε κύριε Χάμπορ, μόλις τώρα το είπατε. Αυτό κατανόησα εγώ. Αυτή ήταν η ενδεικτική πρόταση να γίνει αυτό έτσι. Ναι, τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα λέει η κυρία Γκέμφατ. Λοιπόν, αυτό καλά το κατάλαβα, σωστό. Αλλά όπως γνωρίζετε, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και τις θερινές διακοπές που θα ξεκινάνε. Γι' αυτό προθεσμία για την κατα... κατάθεση τροπολογιών 9η Σεπτεμβρίου είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Παρακαλώ να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, να τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα. Να σας πω και γιατί. Διότι εχθέ στην ομάδα εργασία, όταν συζητήσαμε αυτά τα πράγματα χθε και ανέφερα εγώ αυτά τα οποία είπατε, ποια προσέγγιση ακολουθούμε και ποια χρονοτροχία αρκετοί συνάδελφοι από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είπαν επειδή δεν έχουν εξοικειωθεί σε αυτή τη συζήτηση σε λεπτομέρειες και δεν παρακολουθούν τις συζητήσεις όπως εμείς καθημερινά από πρώτο χέρι, είπαν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι ότι αυτή η νέα προσέγγιση σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα θέματα σε βάθος και σε λεπτομέρειες και πάλι να κάνουμε μια ακρόαση για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας διαφορετικής προσέγγισης ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της δικής σας πρότασης κύριε Σουάμπ εναντί αυτών που είχαμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα και είχαμε δεχθεί. Γι' αυτό δεν είναι καλό στις 9 Σεπτεμβρίου ήδη να έχουμε τελεσίδικα την άποψή μας που θα καθορίσουμε γραπτός διότι στην ομάδα μας τουλάχιστον δεν μας δίνει αυτό τη δυνατότητα να συζητηθούν επαρκώς τα πράγματα, επαρκώς το τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό θα παρακαλούσα θερμά σε αυτή τη διορία, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών να το ξανασκεφτείτε το θέμα και να ξαναπροβληματιστούμε να δούμε ότι για την καλύτερη κατανόηση αυτών που προτείνεται χρειάζεται περισσότερος χρόνος χρειάζεται μια μικρή ακρόαση που θα πρέπει να γίνει πρώτα, ώστε οι διαφορετικές πτυχές να μπορέσουν να φωτιστούν και οι επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν. Στη συνολική προσέγγιση, νέα προσέγγιση που ακολουθούμε τώρα πλέον, γιατί εδώ έχουμε πολλά μπροστά μας που ρυθμίζονται με αυτή την ομοθεσία και αυτές τις προτάσεις. Πρόκειται για την ίδια την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική οι πολίτες οι ίδιοι πρέπει να μπορέσουν να δεχθούν, να μπορούν να δεχθούν αυτά τα οποία κάνουμε εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήταν πολύ αρνητικό αν από παραδρομή, εκ παραδρομής ε, δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε να τους πείσουμε. Κάτι να έχουμε ξεχάσει, κάτι να έχουμε διατυπώσει λάθος και μετά οι πολίτες μετά να μην έχουν εμπιστοσύνη και να δουν ότι αυτό το δικαίωμα, τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν έχουν διασφαλιστεί. Ας πάρουμε περισσότερο χρόνο, μια και έχουμε μια τελείως νέα βάση τώρα ρύθμισης των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέπχαρτ. Είμαι βέβαιος ότι και άλλοι θα θελήσουν να σχολιάσουν το θέμα του χρόνου. Απλώς θεώρησα πως ήταν χρήσιμο να σας αναφέρω τι μας προτάθηκε, αλλά από την Επιτροπή εξαρτάται να αποφασίσει. Και οι θα πρέπει να το σχολιάσει και φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο για τη συζήτησή μας, γιατί είναι σαφές ότι υπάρχουν θέματα που δεν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε Τελείω σήμερα και στι 23 του Ιουνίου μπορεί να χρειαστεί να συζητήσουμε περαιτέρω τα 1, 2, 3 και τα 4, 5. Και Ζώσφορντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Αντρέα, ήθελα ειλικρινά να σα συγχαρώ για την δουλειά σα. Ε, συχνά ε, φαίνεται να είναι τυπική αυτή η διατύπωση, όμως σήμερα ειλικρινά σας συγχαίρω, διότι το κείμενο αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο, εξαιρετικά κακό εξ αρχής και εσείς το δουλεύετε ε, σε βάθος. Κάτι που είναι πολύ επίσης ε, προς τιμή σας είναι ότι κάνετε αυτό που είπατε ότι θα κάνετε. Το πρόγραμμά σας που μας αναφέρατε την πρώτη συνεδρίαση επί του θέματος είναι ακριβώς αυτό που ακολουθείτε. Είναι πολύ ουσιαστική η δουλειά σας και ειλικρινά και πλήρως σας συγχαίρω γι' αυτό. Ε, εσείς επιφέρετε βελτιώσεις πολύ σημαντικές για πολλά ζητήματα συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που μπορεί να φαίνονται καταρχήν επαφανειακά ή όχι για το ουσιαστικά για τους ορισμούς, ας πούμε για το συμβόλαιο πώληση και πραγματικά επιφέρεται μια μεγάλη βελτίωση. Πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα να το βελτιώσουμε, ας πούμε, στα ε, εξ αποστάσεως πωλήσει για την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να βάλουμε στο άρθρο 2 αυτό που βάζετε στο εκτιμώντας 16, δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες της, της βιώσιμης στήριξης. Εν πάση περιπτώσει δύο λεπτομέρειες για να σας αποδείξω ότι και εγώ έχω δουλέψει μέχρι αργά το βράδυ εχθές, το διάβασα, το, το πήρα εχθές το μεσημέρι. Και εγώ. Το βασικό είναι λοιπόν η maximum εναρμόνιση. Και στην ουσία αυτό που προσπαθείτε να κάνετε, αλλά όχι ω ταχυδακτηλουργό, αλλά ω πραγματικό πολιτικό, είναι να διατηρήσετε αυτή την ιδέα τη μέγιστη εναρμόνιση που πολύ άσχημα ξεκίνησε, δίνοντα όμω ένα πεδίο ρεαλιστικό, ένα πεδίο εφαρμογή ρεαλιστικό και εκεί όταν θα έχουμε όλο το κείμενο θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσο το καταφέραμε. Για την ώρα θα έλεγα ότι βρίσκεστε στη μέση ε, και πολύ καλά τα καταφέρνετε και το κάνετε πώς, με εξαιρετικά απλό τρόπο και πρέπει μεταξύ μας να τα λέμε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε, ότι τελικά καταλήγεται δηλαδή σε ένα κείμενο το οποίο όπως έχει τροποποιηθεί δεν είναι πια ένα κείμενο που αφορά μόνο τις πωλήσει ε, εξ ή τις πωλήσει εκτός του καταστήματος. Μιλάμε για μια οδηγία που κάλυπτε σίγουρα αυτά τα σημεία, αλλά που ε, στην ουσία κάλυπτε ένα πεδίο πολύ πιο ευρύ, ενώ εδώ εσείς επικεντρώνετε και πάλι την προσοχή σε, αυτές, σε, αυτό, σε αυτό το θέμα. Εξ αρχής στον τίτλο μιλάτε για στοχευμένη εναρμόνιση. Έχετε δίκιο που υποδεικνύεται ότι στις περιπτώσεις όπου απομένουν, ε, παραμένουν, αποκλίνουν στις εθνικές διατάξεις θα πρέπει τα κρατημέλη να τα κοινοποιήσουν όλα αυτά στην Κομισιόν ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ε, που κατευθυνόμαστε. Δίκιο έχετε επίσης όταν διευκρινίζετε ότι όταν πρέπει να διαρθρωθούν αυτές οι νομοθετικές διατάξεις με άλλες διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται σε άλλα κείμενα προηγούμενα, τα προηγούμενα θα υπερισχύσουν γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξουν αντιθέσεις. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο όλο αυτό θα καλύψει κάθε κίνδυνο αμφισβήτησης. Πάντω ότι το αναφέρετε είναι ήδη πολύ βασικό. Φυσικά παραμένουν κάποια προβλήματα και εδώ στην πρώτη βάθος εξέταση τη, του κειμένου σας έχουμε το εξής πρόβλημα. Στο δίκαιο ανάκλησης αναφέρεται ότι για ε, πολλές χώρες τελειώνει το δικαίωμα αυτό μόλις περάσουν 14 μέρες. Ε, ε, στη χώρα μου αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Ωστόσο μιλήσατε προηγουμένως για τον τεχνίτη που έρχεται στο σπίτι σας για να διορθώσει την μπανιέρα που έχει διαρροή και αυτό μπορεί να είναι θέμα μιας υπηρεσίας ε, όπου μπορεί αυτό να μην ισχύσει και επεξηγείται ότι ο καταναλωτής ε, να γνωρίζει ότι εγκαταλείπει το δικαίωμα ανάκλησης ή υπαναχώρησης. Αυτό δεν είναι πολύ ε, ξεκάθαρο στο κείμενο. Στο άρθρο 19, στο εδάφιο Α, όπου αναφέρεστε όταν μιλάτε για τον τεχνίτη. Το άρθρο αυτό είναι κάπω ε, υπερβολικά όριστο. Θα ήθελα περαιτέρω να το διευκρινίσουμε. Γιατί ω έχει αφήνει να πιστέψει κανεί ότι ο καταναλωτή από τη στιγμή που δίνει τη σύμφωνη του γνώμη αρκεί να δώσει τη σύμφωνη, συμφωνία του, τη σύμφωνη του γνώμη, ώστε τελικά να εγκαταλείψει το δικαίωμα ανάκλησης. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, στο άρθρο 12, εδάφιο 4, ένα πολύ σημαντικό θέμα, λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν στα μέρη να ασκήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καλά τη διάρκεια της ανάκλησης. Στην Γαλλία είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί για πωλήσει εκτός καταστήματος απαγορεύεται να ισχύσουν οι όροι της σύμβασης κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ανάκλησης. Εγώ λοιπόν βρίσκομαι σε μια κατάσταση που για την ώρα δεν με αφήνει να σας ακολουθήσω απόλυτα και το λέτε εξάλλου και εσείς ο ίδιος στο εκτιμώντας 14 όπου εξηγείτε πως πρόκειται τελικά για τις πωλήσει εκτός καταστήματος. Οι πωλήσει εξ αποστάσεων είναι κάτι διαφορετικό, αλλά οι πωλήσει εκτός καταστήματος είναι όταν οι πολιτές πάνε στην κατοικία του καταναλωτή και εξηγείται και εσείς ο ίδιος στο 14 και επαναλαμβάνετε εδώ το αρχικό κείμενο της Κομισιόν με περισσότερες διευκρινήσεις ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση. Όταν δηλαδή ο πολιτής είναι στην κατοικία του καταναλωτή και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γνωρίζουμε πολύ καλά πως για παράδειγμα ο καταναλωτής δεν έχει τα μέσα να συγκρίνει ε, τιμές και αγαθά εκείνη τη στιγμή. Όταν έρχεται ο πολιτής και του προτείνει κάτι στο σπίτι του, πολύ δύσκολο είναι για αυτόν να συγκρίνει τιμές. Και καταλήγουμε σε ένα άλλο προβληματισμό, δηλαδή αρκεί να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκληση, δηλαδή στέλνοντας πίσω το προϊόν, ενώ έχει ήδη πληρώσει και η παράδοση του προϊόντος γίνεται κατά τη διάρκεια τη ίδια της προθεσμίας ανάκλησης. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά, διότι αν υπάρξει κάποια τροποποίηση, Κατά την άποψή μου θα υπήρχε υπαναχώρηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά την εσωτερική αγορά σήμερα, για αυτό το σημείο θα πρέπει να βάλουμε έναν επιταχυντή. Δηλαδή αυτό που είναι ένας μοχλός για την ανάπτυξη είναι οι εξαποστάσεις πωλήσει, δηλαδή οι πωλήσει μέσω ίντερνετ, όπου αρκεί κανείς να κάνει ένα κλικ και αμέσως μπορεί να συγκρίνει τιμές και προϊόντα. Αντιθέτως, στις πωλήσει κατοίκων δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ. Και εδώ αγαπητέ Ανδρέας, διερωτήθηκα τι σας οδήγησε στο να απλοποιήσετε σε τέτοιο βαθμό το άρθρο 10 που μόλις αναφέρθηκε. Εδώ καταργείται ξαφνικά ε, διάφορα τα οποία θα πρέπει νομίζω να επαναξετάσουμε. Για παράδειγμα λέτε ότι με βάση τη φύση της σύμβασης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5. Εδώ ομολογώ ότι πολύ διαρωτώμε, γιατί ούτως ή άλλως όμως θα το μελετήσουμε μέσω των τροπολογιών που θα υποβάλουμε. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί το κείμενο αυτό το λάβαμε χτες αργά και Εν πάση περιπτώσει, από την επιφύλαξη μια πρώτη ανάγνωση που ελπίζω ότι θα σα έπεισα πω το έκανα προσεκτικά, ε, και βέβαια θα πρέπει να εμβαθύνω και περισσότερο. Ε, θα σας πω και περισσότερα σχόλια. Γιατί ο χρονοδιάγραμμα είμαι υπέρ του να καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο από την 9η Σεπτεμβρίου. Αν και ξέρω ότι ήδη αυτό έχει αναβληθεί. Αλλά δεν πρέπει να παγιδευτούμε όπως παγιδευτήκαμε για διάφορα άλλα θέματα. Δηλαδή, αν αναβάλουμε την προθεσμία και κατά συνέπεια καθυστερήσει και η μετάφραση. Αλλά μετά δεν έχουμε πια χρόνο για να δουλέψουμε στο κείμενο γιατί οι μεταφράσεις στάσαν πολύ αργά. Ε, τότε δεν έχει νόημα. Ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να το καθυστερήσουμε. Όχι μόνο ένα στάδιο για να μην μπορούμε μετά να δουλέψουμε με την ησυχία μας για τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό που πιστεύω πραγματικά είναι ότι σε αυτό το κείμενο έχουμε και το βλέπουμε πολύ καλά, όλοι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και χρειάζεται να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και να βελτιώσουμε από κοινού το κείμενο, να προσπαθήσουμε πραγματικά να βρούμε συμβιβαστικέ λύσει και κυρίω στοιχεία συνένεση. και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε το χρόνο όχι μόνο για την κατάθεση των τροπολογιών αλλά και από τη στιγμή που θα έχουμε τη μετάφραση να μπορούμε να δουλέψουμε την ησυχία μα. Και πάλι τελευταία φορά να σα συγχαρώ χαρώ γιατί μπορώ να σας πω ότι με αυτό το κείμενο σήμερα ήδη έχουμε προχωρήσει. Uh, Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κύριε Ροσφόρ. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το χρόνο σήμερα. Προφανώς αυτό δείχνει ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Έχουμε και την κυρία Βόλης που παίζει ρόλο στην νομική επιτροπή και γνωρίζω ότι πρέπει να φύγει για την ψηφοφορία στις 10. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Γουόλης ε, και στους σκιώδεις εισηγητές ε, και μετά θα περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Και δυστυχώς θα πρέπει να βιαστούμε πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή έχω 7 άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είστε πολύ σύντομοι και μάλλον θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα με τον εισηγητή για να αποκτήσουμε μία δομή που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε πολλά θέματα στις λεπτομέρειές τους. Γιατί όπως είπαν πολλοί, οι λεπτομέρειες είναι οι σημαντικές σε αυτό το θέμα. Το λόγο έχει κυρία Βόλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Με συγχωρείτε που θα φύγω, αλλά έχω άλλη συνεδρίαση, πρέπει να μιλήσω αργότερα. Επίσης να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή σας άρχισα να ελπίζω ότι παρέμενα μέλος στην Επιτροπή σας, αλλά βεβαίως ε, όλοι πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφό του και για τις πολύχρωμες διαφάνειες ε, που μας βοηθούν να διαπιστώσουμε τη μεθοδολογία που σκοπεύει να ακολουθήσει. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ανησυχεί κατά βάση για το πώς θα βρούμε ένα τρόπο έτσι ώστε αυτή η οδηγία να συνεργαστεί καλά με οποιαδήποτε πρόταση προκύψει από το έργο που γίνεται για το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συμβάσεων, που αυτή την περίοδο προχωράει καλά συνεκλήθη για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα μία Επιτροπή Εθνικών Εμπειρογνωμόνων η οποία θα έχει στη διάθεσή της ένα έτος για να καταλήξει στα 150 περίπου άρθρα ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο που ενδεχομένως, ενδεχομένως να γίνει προαιρετικό δεσμευτικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσαν να εγκρίνουν επιχειρήσεις δημιουργώντας ένα τύπο ενοχικού δικαίου υπεράνω του εθνικού δικαίου. Και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βελτιώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Επαναλαμβάνω, αυτό θα είναι προαιρετικό, ενώ εδώ η οδηγία για τους καταναλωτές θα είναι υποχρεωτική. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι πρόκειται για δύο εναλλακτικές λύσεις εδώ. Εγώ όμως θεωρώ ότι μπορούν να συνεπάρξουν. Και τώρα που είδα και την παρουσίαση του κυρίου Σβάμπ, παραμένω πεπισμένη για αυτή τη δυνατότητα συνύπαρξης. Γι' αυτό όμως το λόγο πρέπει να είναι πολύ σύναφη μεταξύ τους. Πρέπει να κινηθούμε λοιπόν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πολλοί από τους προλαλήσαντες ανέφεραν λεπτομέρειες που θα εξετάσουμε. Γιατί όλοι θα βρουν κάποιες λεπτομέρειες που διαφωνούν με τις εθνικές τους ρυθμίσεις και που ίσως φαίνονται ότι μειώνουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όσο λοιπόν πιο πολλές τέτοιου είδου διαφορές ε, εμφανίζονται, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Εμείς πάντως στη Νομική Επιτροπή έχουμε πολλά προβλήματα με χρονοχρονά διάγραμμα, γιατί θα πρέπει να προηγηθούμε της δικής σας επιτροπής για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε γνωμοδότηση και επίσης εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα και εγώ όπως και άλλοι να ζητήσω λίγο παραπάνω χρόνο. Πρόκειται για θέμα που έχει μείνει στα συρτάρια μας για πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται τώρα να βιαστούμε. Το σημαντικό είναι να βγάλουμε κάτι ορθό, καλό. Είναι πολύ σημαντικές οι λεπτομέρειες και η συνέφεια με το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε για την πολύ καλή αρχή. Αναμένουμε με ανυπομονησία τις περαιτέρω συζητήσεις, αλλά παρακαλούμε λίγο παραπάνω χρόνο. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε και για την μεγάλη δέσμευσή σας. Όσον αφορά τις διαδικασίες, προφανώς αυτό το θέμα θα πρέπει να το συζητήσει ο εισηγητής με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και μέσα από την Νομική Επιτροπή. Είχαμε μία συμφωνία, αλλά ίσως θα έπρεπε να την αναθεωρήσουμε αν υπάρξουν εξελίξεις ε, στο κεφάλαιο 5, που αφορούν ε, την νομική επιτροπή. Εσείς λοιπόν μαζί με τον εισηγητή μας θα πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα και ενδεχομένως να επαναξιολογήσετε τα, τους κανόνες που θα ισχύουν για την ανάμειξή σας. Τώρα, η κυρία Τσούρνεν εκ μέρους ε, των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περιμένω όλοι να βάλουν τα ακουστικά τους. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το δημιουργικό του έργο. Να πω και στην κυρία Γκέμπχαρντ ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω αυτή την επιλογή χρωμάτων κόκκινο και πράσινο. Να πω πάντως κάτι στη γραμματεία. Όταν λαμβάνουμε ένα κείμενο αργά το βράδυ, αυτό περιπλέκει πολύ τα πράγματα. Εγώ έλαβα το κείμενο χτες στις 5 παρα 20. Προσπάθησα να το διαβάσω χτες το βράδυ, αλλά δουλεύαμε και όλη την ημέρα χτες. Δεν βοηθάει αυτό αν θέλουμε να έχουμε επικοδομητική συζήτηση. Θα θέλαμε λοιπόν να λαμβάνουμε τα έγγραφα νωρίτερα. Ένα αυτό. Περνάω όμως τώρα σε κάποια ερωτήματα. Ως σκιώδη συζητήτρια μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα και διμερός. Όμως, αν εδώ μιλάμε για μία ομπρέλα που θα καλύπτει πολλά πράγματα για τους καταναλωτές ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάποιες επιλογές. Ελάχιστες ή μέγιστες προϋποθέσεις. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες αμφιβολίες για την επιλογή που κάνατε εσείς. Και βλέπω ότι χρησιμοποιείτε ένα διπλό μοντέλο που δεν είμαι σίγουρη ότι αυξάνει την νομική ασφάλεια. Αν θέλουμε νομική ασφάλεια, πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Το σύστημα που προτείνεται αναρωτιέμαι μήπως είναι υπερβολικά περίπλοκο για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Βλέπω και στη Δανία ότι οι επιχειρήσεις αρχικά ήταν πολύ ικανοποιημένε, αλλά τώρα έχουν πολλές αμφιβολίες γιατί δεν είναι αρκετά σαφές το κείμενο. Βεβαίως ε, τελικά ίσως το κείμενο του κυρίου Σβάμπ να είναι πιο σαφές από την πρόταση αυτή καθ' αυτή της Κομισιόν. Γιατί όντως αυτό που πρέπει να δούμε είναι το πόση εναρμόνιση χρειαζόμαστε σε κάθε κεφάλαιο. Να πω επίσης ότι συμφωνώ απολύτως με την κυρία Γουόλης που μίλησε για την σχέση εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για τις συμβάσεις. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προκειμένου να μην έχουμε ένα υπερβολικά δυσανάγνωστο μείγμα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα, ναι, χρειαζόμαστε χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να, να αναβάλουμε την απόφαση. Και σίγουρα θα έχουμε και χρόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών να μελετήσουμε το θέμα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία παράταση στην προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Τούρναν. Πολύ σύντομα να μιλήσω και εγώ ως σκιώδης συζητήτη του ECR. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ανδρέας γιατί κατέγραψε σαφώς τη στρατηγική που επιθυμεί να ακολουθήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντική αλλαγή σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Βέβαια, η νέα Επιτροπός, η κυρία Ρέντινγκ, μας λέει ότι μάλλον είναι πιο θετική. Άρα, ίσως ε, κινηθούμε όλοι προς μια κοινή κατεύθυνση όσον αφορά τη δομή. Και από ό,τι φαίνεται και το Συμβούλιο πρόκειται να συμφωνήσει. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ένα ενοποιημένο κείμενο εφόσον πρόκειται για πολύ πολύπλοκη πρόταση. Βεβαίως, όπως είπε και η κυρία Κέπχαρτ, θα χρειαστεί να δούμε το κείμενο στο σύνολό του για να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ασαφίες ή αμφισημίες ε, τις λεπτομέρειες. και υπάρχουν και θέματα που προκύπτουν από την προσπάθεια τροποποίησης άλλων οδηγιών, για παράδειγμα της οδηγίας για τις πωλήσει εξ αποστάσεων. Σίγουρα όμως η νέα δομή είναι πολύ πιο λογική, πολύ πιο καθαρή, αλλά όπως υπόθηκε όλοι θα χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Τώρα όσον αφορά τα πολύχρωμα διαγράμματα. Κοιτάξτε, στα κεφάλαια 4 και 5 έχετε λίγο κίτρινο στο μέσο, αλλά εγώ νομίζω ότι είτε θα έχουμε εναρμόνιση, πράσινο εκεί, είτε όχι. Το σημαντικό είναι ότι όπου θα έχουμε εναρμόνιση θα έχουμε κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για τους καταναλωτές που θα είναι απαραίτητες και στα 27 κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει εναρμόνιση και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Εσείς μας λέτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε πλήρη εναρμόνιση, σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να προσθέσουν επιπλέον προϋποθέσεις. Το πολύ σημαντικό όμως εδώ είναι οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές. Τέλος, και θα ήθελα να δω αν συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου, υποθέτω ότι αυτό είναι κομμάτι μιας ε, διαρθρωμένης προσέγγισης της Κομισιόν για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Οι πίτροποι Ρέντιν και Ντέλη ασχολούνται με τις διαφορετικές διαστάσεις και αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε είναι να υπάρξει συντονισμός όλων αυτών. Τώρα, λέτε σε κώδικα πάγωμα και αξιολόγηση ομοτήμων. Υποθέτω ότι αυτό που εννοείται είναι ότι αν εγκριθεί αυτή η οδηγία, δεν θα πρέπει να υπάρξουν νέες διατάξεις που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό των οδηγών. Θα έχουμε λοιπόν μια στατική οδηγία και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε το τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό πάντως είναι κάτι το πολιτικό που θα πρέπει να το συζητήσουμε ως πολιτική επιλογή. Τώρα, όσον αφορά την ε, επικοινωνία. Έχουμε συζητήσει με την Κομισιόν για την οδηγία για τους καταναλωτές και τη μεταφορά τους. Κύριε Μάντερς, παρακαλώ. Τουάν. Λοιπόν, στην οδηγία για τη καταναλωτική πίστη είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι αυτή η οδηγία θα συνδέεται απρόσκοπτα με την οδηγία για τους καταναλωτές. Και εφόσον η οδηγία για την καταναλωτική πίστη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία, πρέπει να, να προσέξουμε πολύ αυτό το θέμα. Και σας υπενθυμίζω ότι πολλές από τις διατάξεις ε, της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη αφορούσαν τα καταναλωτικά δάνεια κτλ. Που βεβαίως πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υπάρχουν ασυνάφειες μεταξύ των δύο. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Τριανταφυλλίδης παρακαλώ. Δεν σας βλέπω πολύ καλά, αλλά παρακαλώ έχετε το λόγο. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Άντρεας για την εξαιρετική δουλειά που έχει παρουσιάσει και τον συγχαίρω Είχαμε ως κοιόδης συζητητές ε, αρκετές συναντήσεις μαζί του. Μας εξήγησε την αρχιτεκτονική που θα ακολουθούσε και τώρα που είδα τις ε, διαφάνειες έχω αντιληφθεί πλήρως το στόχο που επιδίωκε που ήταν να βρει μια λύση με την πλήρη εναρμόνιση εκεί όπου χρειαζόταν ε, και κάτι άλλο εκεί που δεν μπορούσε να γίνει πλήρης εναρμόνισης. Επομένως, αυτή η ιδέα της αμπρέλας πιθανόν να πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, σε ό,τι αφορά τα, κάποια σημεία που είχαμε ε, διαφορετική άποψη στο παρελθόν, δεν ξέρω αν καλύπτονται από το έγγραφο που έχει παρουσιαστεί, αλλά θα συμφωνούσα με αυτό που είπε η κυρία Γκέμπαρτ προηγουμένως, ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποβαθμιστεί η προστασία του καταναλωτή και δυστυχώς αν παραμένει η αναφορά που υπήρχε ότι η στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση δεν πρέπει να μειώσει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών, εμείς διαφωνούμε γιατί ασφαλώς δεν πρέπει να μειώσει καθόλου, όχι να μειώσει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, ε, ε, το γεγονός ότι δεν καλύπτονται συναλλαγές από επιχείρηση σε επιχείρηση το θεωρούμε σαν μια δυναμία. Οι κοινοί ορισμοί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά πρέπει να εξαλειφθούν κάποιες αποφάσεις που υπάρχουν. Στο θέμα των τιμών ε, πρέπει να γίνει σαφές ότι ο καταναλωτής γνωρίζει την τιμή και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να είναι καθαρό ε, αυτό το ζήτημα ε, συμφωνούμε με τον καθορισμό των 14 ημερών, αλλά πρέπει να διασαφανιστεί ότι η περίοδος υπαναχώρησης θα πρέπει να ισχύει από την περίοδο ε, παραλαβής του προϊόντος και όχι από τη στιγμή που στέλνεται το έντυπο παραγγελίας. Ε, επομένως πρέπει να εξετάσουμε αυτό το, αυτές τις λεπτομέρειες στο έγγραφο και να επανέλθουμε. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα έχει σχολιαστεί επαρκώς. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο περισσότερο χρόνος και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θα κάνουμε τώρα λοιπόν, αν συμφωνείτε και οι υπόλοιποι, είναι να διακόψουμε τη συζήτηση. Να ψηφίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και μετά να δούμε και τον χρόνο των υπόλοιπων ομιλητών, γιατί φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούσετε και την Κομισιόν και το Συμβούλιο και τον εισηγητή. Κοιτάω, ναι, θα θέλατε να έχετε σχόλιο από πλευρά τη Κομισιόν και Συμβουλίου. Ίσως να μην προλάβουμε να ακούσουμε όλους τους ομιλητές σήμερα, αλλά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αν δεν προλάβουμε. Λοιπόν, ψηφοφορία. Δεν πρότεινα να ψηφίσουμε με τις κάρτες σήμερα γιατί νομίζω όμως ότι τελικά θα μπορεί και να τις χρειαστούμε, μπορεί και όχι. Well, at the moment, we, my plan is not to vote with cards, so let's uh, proceed. Now, the first uh, proposal is the um, draft opinion from Mr. Fox. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση του κ. Fox για τα δίκαια εισοδήματα των uh, γεωργών. Παρακαλώ, όσοι αποχωρείτε, ησύχως. Και να μην κουβεντιάζετε όσο ψηφίζουμε, παρακαλώ. Κύριε Φόξ, θέλετε να πείτε τίποτα πριν την ψηφοφορία. I want to, uh, thank you very much for your energetic work as in Σας ευχαριστώ πολύ γιατί ως εισηγητής μπορέσατε να ξεκαθαρίσετε διάφορες, συμβιβα... διάφορες τροπολογίες, να κάνετε συμβαστικέ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Ψηφίζουμε λοιπόν για την πρόταση του κυρίου Φόξ. Είστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσετε. Ωραία. Να ψηφίσουμε πρώτα για τη συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παγιωμένη 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 6. Ζουβέν Σβάμπ Μπίλτ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 10. Ζουβά και Κοράτσα Μπίλτ. Με προφορική ε, τροπολογία που έχει δημοσιευθεί. Υπέρ με την προφορική κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Φόξ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ζουβά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παγιωμένη τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Με προφορική ερώτηση που την έχετε του κυρίου Ζουβά. Υπέρ κατά. Νομίζω πως εγκρίνεται. Μπορείτε να ξανασηκώσετε τα χέρια σας. Υπέρ, ποιοι είναι, παρακαλώ. Twenty-two in favour. Mm-hmm. Can we check the numbers of the EPP? Those against. Kata. How much? 13, okay. So that, that is carried. What was the number? 22 in favor and 13 again. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τρία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 17. Υπέρ. Υπέρ για να μετρήσω παρακαλώ.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 κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική, μάλλον στην τροπολογία 21, Ζουβά έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 22 τώρα, του κυρίου Ζουβά, υπέρ. 22 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Δεν σα είδα εκεί πέρα που υπερψηφίσατε την ίδια σας τροπολογία. Κάποιον έψαχνα υπέρ. Τροπολογία 23 του κυρίου Ζουβά. 5 υπέρ. Κατά. Οι υπόλοιποι κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 28 του κύριου Φόξ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 29 με προφορική τροπολογία που είναι εδώ, ε, την έχετε δει, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, φόξ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η παγιωμένη 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στην 33, του κύριου Φόξ και της κυρίας Βέστφαλ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. Και έτσι πάμε στην 34 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. 35 Ζουβά υπέρ. Πάλι πρέπει να μετρήσουμε. 35 ποιοι είναι υπέρ.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 19 uh, um, against. 19 κατά, οπότε απορρίπτεται. 18 υπέρ, 19 κατά. 36 Ζουβά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και έτσι τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης και πρέπει να μετρήσουμε υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε ομόφωνα λοιπόν. Μπράβο κύριε Φόξ και ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν η πρώτη σας νομοδότηση για την Επιτροπή ή η δεύτερη. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Uh, the report from Louis Grech, uh, who unfortunately I know is not able to be here, but I think Mrs. Uh, Gephardt will stand in for him if we have any queries, but I think we can just go ahead with the vote. Πάμε στην έκθεση ψήφιση της εκθέσης Grech, που δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε εδώ μια γνωμοδότηση για τις εφαρμοστικές διατάξεις της Κομισιόν, αρμοδιότητες μάλλον της Κομισιόν. Ε, το ξεκινάμε. Πρώτη τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. Ήταν η 4. Η 9. Γκρέχ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 5, 6 και 7 θεωρούνται πως ε, εγκρίνονται ε, μαζί με την 9. Έχουμε τη 19. Μπουζόη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 γκρέχ υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 10, γκρέχ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 11, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία 20 με προφορική τροπολογία μπουζόη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 καταπίπτει και πάμε τώρα στη 13 γκρέχ υπέρ. όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Η 13 απορρίπτεται. Και αυτή πάμε τώρα στο άρθρο 9. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε on block, αυτές που αφορούν το άρθρο 9, οι δύο δηλαδή, 21 και 22. Υπέρ ποιοι είναι. Α, όχι. Συγγνώμη. 21, ναι. 21, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, άρα η 22 καταπίπτει. Και περνάμε στις τροπολογίες 23 και 24, τις οποίες μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Πάμε τώρα στην ε, εκτιμώντας. Έχουμε τροπολογία 1, γκρέχ, ποιοι είναι υπέρ, κατά ε, εγκρίνεται 2 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 16 με προφορική τροπολογία μπουζόη ποιοι είναι υπέρ κατά εγκρίνεται η τροπολογία 17 υπέρ κατά εγκρίνεται η 18 καταπίπτει και ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης όπως το υπέρ Κατά εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Λουί Γκρέσ παρότι λείπει. Και τελευταία ψηφοφορία είναι για την κυρία Σούγη. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Σούγη. Θέλετε κάτι να πείτε πριν από την ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλα έχουν πάει πολύ καλά και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν εδώ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Προχωράμε λοιπόν στην γνωμοδότηση της κυρίας Σούλη. 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 η Κορέα Ντεκάμπος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 με προφορική τροπολογία που την έχετε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Κορέα Campos. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 με προφορική του Ντιγιόν Kreutzmann υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 10 σουγή υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 14 υπέρ κατά εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 με προφορική ε, ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 17 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 18 με προφορική τροπολογία Κορέα Campos υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας, εκτιμώντας α, προφορική τροπολογία σουγή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. 3 έχει αποσυρθεί, τροπολογία 4 με προφορική υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και το σύνολο της γνωμοδότησης τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σουγή για την πρώτη σας νομοδότηση. Ελπίζω να υπάρξουν και πολλές άλλες. Έτσι κλείνουμε με τις ψηφοφορίες, τελειώσαμε και αυτό που προτείνω είναι να συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση την τόσο σημαντική του κυρίου Σοβάμπα. Πρέπει να έχουμε τελειώσει γύρω στις 11, γιατί ο κύριος Ζουβά τότε θα μας παρουσιάσει τη δική του έκθεση, ίδιας πρωτοβουλίας. Να κάνω την εξής πρόταση, να τσεκάρω ποιους έχω εδώ ε, ως ομιλητές, να δω αν θέλει κανείς να προσθεθεί. Mrs. Mr. Correa uh, and Mr. Kreutzmann. Uh, So that's one, two, three, four, five, six, seven speakers. Anybody else want to contribute? Uh, Then uh, Ms. Aris has to leave, so that we have uh, one, two, three, four, five, six. Uh, Then I'd like to hear from Mr. Pronk and Mr. Crespo. Um, Would... uh... Και μετά θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Πρόν και τον κύριο Κρέσπο. Θα ήθελα τότε να σας καλέσω, α, ναι, και τον κύριο Σβάμπ στο τέλος, Παρακαλώ λοιπόν δύο λεπτά να πούμε για τον κάθε ε, ομιλητή. το δέχεστε. Ωραία λοιπόν. Να δώσω στην Αντιπρόεδρο Μπερνιέ το λόγο για, δι... Βερνιό, για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήδη έχουν υποθεί αρκετά να ευχαριστήσω τον κύριο Σβάμπ που για το προσεκτικό του έργο που βεβαίως τώρα μόλις αρχίζει. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε τις συζητήσεις ε, και σε μία συνεδρίαση υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας. Τώρα, για τις λεπτομέρειες. Να πω ότι η κυρία Ρέντινγκ είναι λιγότερο ευνοϊκή στην πλήρη εναρμόνιση που αυτή τη στιγμή μου φαίνεται απίθανη. Όμως, ένα σημείο στο οποίο πρέπει να έχουμε πλήρη εναρμόνιση, κύριε Σφάμπ, είναι στο δικαίωμα υπαναχώρησης. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και σε άλλες οδηγίες που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών Πρέπει λοιπόν να έχουμε στόχο 14 ημέρες ε, δικαίωμα υπαναχώρησης για όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Μετά, για τις λεπτομέρειες. Είπατε ότι όντως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες ε, που έχουν πρόβλημα. Είχαμε και μία μελέτη πρόσφατα αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία που έδειξε πόσο πολλές απέ... απάτες υπάρχουν εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε οι πολύ ευάλωτοι καταναλωτές πέφτουν θύματα απάτης, πραγματικής απάτης. Και εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του δικαιώματος του καταναλωτή για τις ε, τραπεζικές υπηρεσίες το οποίο θα, θα προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή στις, στους όρους παροχής των υπηρεσιών χωρίς γραπτή έγκριση από τον καταναλώτη. Κάθε φορά που ο καταναλωτής ανοίγει έναν λογαριασμό, οποιονδήποτε λογαριασμό, πολλές φορές μας τα λένε όλα από το τηλέφωνο, δεν υπογράφουμε τίποτα. Πρόσφατα εμένα μου έτυχε αυτό με μία σύμβαση κινητής τηλεφωνίας. Είχα ζητήσει διάφορα πράγματα από το τηλέφωνο και όταν ήρθε τελικά η σύμβαση περίχε πολλά πράγματα που δεν μου τα είχαν πει από το τηλέφωνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με απάτη. Ένα αυτό. Τώρα όσον αφορά τον χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Ακόμη και αν δουλέψουμε όλο τον Αύγουστο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε σημαντικές ε, τροπολογίες και να βρούμε καλούς συμβιβασμούς με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις τροπολογίες της 9 Σεπτεμβρίου για να συζητηθούν 26 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βιαστούμε γιατί εδώ πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ και αναμένουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε την κυρία Βερνιό. Σας δώσαμε λίγο χρόνο παραπάνω επειδή είστε αντιπρόεδρος. Μπουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου σήμερα για να τα καταφέρω σε δύο λεπτά να τηρήσω τον χρόνο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Και είναι σημαντικό να βρούμε τη σωστή βάση που θα πετύχουμε. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις για κάτι τέτοιο. Αν όμως υπάρχει η πολιτική βούληση αν συμφωνήσουμε στις βασικές θεμελιώδεις αρχές, τότε σίγουρα μπορούμε να βρούμε λύσεις και στις λεπτομέρειες και στα εξειδικευμένα θέματα. Η πρόταση του συναδέφου Σβάμπ είναι πολύ καλοδεχούμενη. Εξαιρετική δουλειά έκανε ο κύριος Σβάμπ, ώστε να καθοριστούν οι κανόνες όσον αφορά έναν απόλυτο πλήρη εναρμονισμό για τις τηλεσυμβάσεις, τηλεπολίσεις, Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές ε, μεταξύ των κρατών μελών. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά κάποιες ε, συμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα προϊόντα, πολύ καλά τα όσα μας είπε. Πρέπει ο καταναλωτής πρώτα να ενημερώνεται για το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ανάκλησης. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν και κυρώσεις μέσα στο πλαίσιο ενός έτους, αν δεν έχουν ενημερωθεί σωστά οι καταναλωτές ανάκληση, περίοδος ανάκλησης σε 14 ημέρες. Καλό αυτό. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις που στην πρακτική εφαρμογή ε, μπορούν να λειτουργήσουν. Θέλω να υποστηρίξω τις προτάσεις. Θέλω να πω όμως ότι ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπάρχει κατάχρηση από πλευράς κάποιων καταναλωτών. Και για τη βιομηχανία δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις που εδώ πρέπει να εισαχθούν για κάποιες ε, προϋποθέσεις. Τότε μπορούμε ένα καλό περίγυρο να διασφαλίσουμε. Την κυρία Γκέπαρντ, ε, τον κύριο Χωσφό και όλους τους άλλους συναδέφους και σκιώδεις εισηγητές ευχαριστώ. Είναι οι επαΐοντες από πλευράς μας αυτοί και οι σκιώδεις εισηγητές έχουν σαφέστερες απόψεις ε, για όλα αυτά τα θέματα επειδή έχουν εξοικειωθεί με τα θέματα. Γνωρίζω τον κύριο Σουάμπ και είμαι έχω τη βεβαιότητα ότι όλες αυτέ οι προτάσεις για βελτίωση θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη. Χαιρετίζω την πρότασή του, την προσέγγιση του συνολικά. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Donc... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα. Καταρχάς, κάτι που είπαν και άλλοι, το χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και δεν πρέπει να βιαστούμε. Λάβαμε χτες ένα περίπλοκο κείμενο και πρέπει σήμερα να κάνουμε την πρώτη συζήτηση. Πολλοί από εμάς δεν προλάβαμε να δούμε το κείμενο. Χρειαζόμαστε χρόνο λοιπόν. Δεύτερο, τι θέλουμε. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ζητούσαμε την μέγιστη δυνατή εναρμόνιση. Εξάλλου, γι' αυτό μιλάμε για οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η αναδιατύπωση ορισμένων διατάξεων από τον κύριο Σφάμπ έχει γίνει πολύ έξυπνα και ρεαλιστικά θεωρώ ότι βρισκόμασταν σε αδιέξοδο, αλλά σιγά σιγά καταφέρνουμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Παρ' όλα αυτά, θα κάνω κάποια σχόλια. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τις ε, νομικές ε, διακριβώσεις ε, για τις συνθήκες πώλησης, τα ευαίσθητα συμβόλαια υπάγονται σε ελάχιστη εναρμόνιση, δεν εξαιρούνται, αυτό είναι θετικό. Τώρα, κάποια πράγματα για τα οποία έχω αμφιβολίες. Άρθρο 5 για παράδειγμα γιατί εκεί μιλάμε για ενημέρωση για τους ε, εμπορικούς κανόνες και τις υπηρεσίες μετά την πώληση. Επίσης, στο άρθρο 11 αναφέρεται αν αυτό θεωρείται κατάλληλο με βάση τη φύση της σύμβασης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό ακριβώς, ίσως να φταίει ότι το διάβασα κείμενο. Στο άρθρο 5 σημείο 3 δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Εν πάση περιπτώσει, το κείμενο περιέχει πρόοδους και περιέχει και διεξόδους αλλά υπάρχουν πολλά ερωτήματα που απομένουν. Όντως υπάρχουν πολλά ερωτήματα και θα πρέπει να βρούμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πάνω, περισσότερο από όλα μια ενημέρωση που σχετίζεται και με τις πληροφορίες ε, για την υπόθεση των, ε, της κλωστοϊφαντουργίας. Όταν αγοράζει κανείς ε, με συγκεκριμένο τρόπο σε ένα κατάστημα και όχι άμεσα στον καταναλωτή, ας πούμε ένα ρούχο, τη στιγμή που μπορεί να αρέσει, να μην αρέσει, μπορεί να είναι ελαττωματικό, έχουμε δυσκολία να καταλάβουμε αν η ευθύνη είναι του διανομέα ή αν είναι του παραγωγού. Θεωρώ λοιπόν πως ήταν σκόπιμο και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στην ε, κλωστή να ξέρουμε αν ο καταναλωτής ε, θα πρέπει να στραφεί στον διανομέα, στον έμπορο δηλαδή, ή αν θα πρέπει να στραφεί στον ε, παραγωγό. Αυτό ισχύει και για ενδεχόμενες αλλεργίες που μπορεί να προκληθούν λόγω του υφάσματος, παραδείγματος χάρη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Στην Ιταλία είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα και προβληματικό. Χρησιμοποιούνται τα διάφορα call center, τα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά δεν λειτουργούν πάντα. Ε, πολύ συχνά είναι προβληματική η κατάσταση. Εγώ να χαρώ και τον Αντρέα και τους σκιώδες εισηγητές γιατί είναι δύσκολο το θέμα και είναι και ευαίσθητο και σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Uh, um, Ευχαριστώ την κυρία Κομή. Κορέγιαντε Κάμπος. Εγώ συμφωνώ με τα σχόλια που ακούστηκαν όσον αφορά την μέθοδο ανάλυσης του Ανδρέα Βάμπα και τους σχετικούς επένου, Ωστόσο, όσο περισσότερο αναλύουμε, τόσο περισσότερες αμφιβολίες έχουμε. Αν κοιτάξουμε αυτό το γράφημα εδώ με τα κυλίνδρους, αυτοί που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 και στο κεφάλαιο 5, έχει μια φράση στο τέλος που λέει το εξή. Λέει, Other dispositions, άλλες διατάξεις ε, θα διατηρηθούν στην αρχική οδηγία και ενώ στους κυλίνδρους που αφορούν το κεφάλαιο 5 λέει ότι άλλες διατάξεις θα παραμένουν στην αρχική οδηγία. Εγώ τι καταλαβαίνω από αυτό, ότι το πρώτο αφορά τις τέσσερις οδηγίες που πρέπει εδώ να συγκεντρωθούν και το δεύτερο αναφέρεται στις ε, οδηγίες από τις οποίες πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις. Το ένα είναι με κεφαλαία γραμμένα, το άλλο είναι με μικρά. Τώρα, για το 4. Άλλες διατάξεις θα διατηρηθούν στις αρχικές οδηγίες, δηλαδή θα διατηρήσουμε τις τέσσερις οδηγίες που θέλουμε εμείς εδώ να τις ε, συγκεντρώσουμε, θα διατηρήσουμε ενισχύ. Άρα δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα σε αυτό. Δεύτερη μου παρατήρηση. Υπάρχει, έχω μια αμφιβολία όσον αφορά τη στοχευμένη εναρμόνιση και είναι η εξή. Σε σχέση με τα όσοι ήδη εδώ συζητήθηκαν, την πρόταση δηλαδή της ε, Επιτρόπου Ρέντινγκ για να ξεχωρίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο από τα υπόλοιπα για να προσπαθήσουμε την πλήρη εναρμόνιση όσο αυτό γίνεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εντάξει, υπάρχουν όμως εδώ δύο αξίες που τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το πρώτο είναι ότι όλοι συμφωνούμε να αναπτυχθεί περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεύτερη αξία είναι ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και συμφωνούμε όλοι από αυτό. Αλλά αυτά τα διέρχονται σε αντίθεση γιατί αν διευρυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο με πλήρη εναρμόνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου περιορίζει το περιθώριο εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει ο καταναλωτής. Από την άλλη πλευρά, συμφωνούμε και δεχτούμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί καλά μέσα σε κάθε κράτος χωριστά, αλλά διασυνοριακά όχι. Με αυτό στην ουσία αφαιρούμε τις προϋποθέσεις ε, πάνω στις οποίες βασίζεται το ηλεκτρικό εμπόριο. Εγώ δεν έχω γνώμη, δεν ξέρω ποια είναι η λύση, αλλά προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Δεύτερο θέμα, καλύτερη προστασία στην ε, κατοίκων πώληση face to face και καλύτερη προστασία στο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια υπηρεσία. Δηλαδή, αντίστοιχα, ανάλογα με το αν ένα αγαθό ή υπηρεσία έχει πολιθεί μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου ή αν έχει πολιθεί πωληθεί face to face, έχει, έχουμε διαφορετική συμπεριφορά και κάλυψη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, αλλά πρέπει να το τονίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους καταναλωτές χρειαζόμαστε πάντα καθαρούς κανόνες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Πρέπει να επικεντρωθούμε επί ορισμένων θεμάτων και κυρίως επί των καθαρών κανόνων. Για παράδειγμα, έχουμε πολλές φορές μη σοβαρούς ε, παραγωγούς οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες άχρηστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει ο καταναλωτής ο οποίος πέφτει στην παγίδα να μπορεί να ξεφύγει από αυτήν, να ξεφύγει από αυτή την απάτη. Στο άρθρο 11 που μιλάτε για παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς ότι απαιτείται σύμβαση ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής ακριβώς επιτίνος συμφωνή και να υπάρχει και σαφής δήλωση από τον καταναλωτή ότι αυτό ζητάει. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλες τις συνέπειες. Είναι πολύ σημαντικό από τη μία πλευρά να προστατεύουμε προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, να αυξήσουμε τα δικαιώματά τους, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι πάροχοι θα γνωρίζουν ότι θα λάβουν πληρωμή για τις υπηρεσίες τους και ότι δεν θα έχουμε συνεχώς επιστροφές προϊόντων, κάτι που θα καταλήγει στον εκμηδενισμό του κέρδους των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία ανεκτή συμβιβαστική λύση, χωρίς να δημιουργήσουμε υπερβολικό άγχος για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Επειδή λείπει ο κύριος Αρίας, θα δώσω το λόγο στην Σουζάνα και θα την αφήσω να μιλήσει αυτή ανταυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε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 Εντάξει, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Να ξεκινήσω ξανά, ναι, ναι. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι στην προηγούμενη θετία είχαμε εγκρίνει μια έκθεση που συμπεριλάμβανε μια κοινή πρόταση με που ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε συμβάσεις modal διαφορετικών τύπων για τις πωλήσει από το διαδίκτυο. Έτσι, οι πολιτές οι οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν σύμβαση διαφορετικού τύπου θα έπρεπε να αναφέρουν σε τι ακριβώς διέφερε το συμβόλαιό τους από τα κλασικά συμβόλαια τα συμβατικά συμβόλαια. Επίσης, είχε συζητηθεί το θέμα της εμπιστοσύνης και το κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους δείκτες εμπιστοσύνης που θα επέτρεπαν στους καταναλωτές να λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις. Μετά υπάρχει το θέμα του κώδικα δεντολογίας. Πολύ σημαντικό και χαίρομαι γιατί ασχολείται με το θέμα η κυρία Ρέντινγκ. Ίσως θα έπρεπε να το δούμε και στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σε μια ώρα έρχεται η κυρία Ρέντινγκ, ίσως θα έπρεπε να θέσετε το θέμα. Ελπίζω να παραμείνετε για να κάνετε αυτή την ερώτηση. Α, συγγνώμη, κυρία Κρούσα έρθει μετά. Έχω αρχίσει να τα μπλέκω. Η κυρία Ρέντινγκ παραμένει επίκαιρη για την Επιτροπή μας, αλλά όχι. Στις 11 η κυρία Κρούς θα έρθει, όχι η κυρία Ρέντιν. Λοιπόν, Μπάρτο για τις συμβάσεις τις καταναλωτικές. Thank you, uh, Chairman. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά τώρα. Καταρχάς να συγχαρούμε τον κύριο Σφάμπ. Μάγνους Όπους έχουμε εδώ. Ένα τεράστιο έργο και συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να εργάζεται κανείς με τόσο πολλές νομοθετικές πράξεις ισχύουσες και ο κύριος Σβάπ σίγουρα έκανε μια επιτυχή προσπάθεια. Και νομίζω ότι ευθυγραμμίστηκε και με τις ανάγκες του Κοινοβουλίου αλλά και με την ομιλία της Επιτρόπου πριν από λίγο καιρό εδώ στην αίθουσά σας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή εκκίνηση της διαδικασίας. Σίγουρα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, εκατοντάδες λεπτομέρειες, σημαντικές για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς θα χρειαστεί πολλή συζήτηση επί των λεπτομεριών αυτών. Όσον αφορά τώρα την ε, αναδιάρθρωση της έκθεσης είναι προφανές ότι επικεντρώνεστε στα πιο σημαντικά θέματα για την εσωτερική αγορά, κάτι που ανέφερε και η ομιλία της Επιτρόπου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συγητής απομακρύνεται από την αρχική πρόταση. Για παράδειγμα, προτείνοντας περίοδο αναμονής ενός έτους αντί για τρεις μήνες. Και υπάρχουν και άλλα θέματα όπου έχουν γίνει αλλαγές που επιδεινώνουν την θέση των καταναλωτών. Επίσης Θεωρείτε ότι το email δεν συμπεριλαμβάνεται στα μόνιμα μέσα, δεν μπορεί δηλαδή να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχάρησης ο καταναλωτής μέσω email. Εν πάση περιπτώσει όμως, κινήστε προς την σωστή κατεύθυνση και θα επαναλάβω αυτό που είχε πει η Επίτροπος είναι σημαντικό να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των παρόχων των υπηρεσιών και των καταναλωτών. Και να μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά παράπονα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί πολλές χώρες εξακολουθούν να μην καλύπτονται καθόλου από επιχειρήσεις, ειδικά στις, ε, στα νέα κράτη-μέλη, αλλά και σε ορισμένα παλαιά μικρότερα κράτη-μέλη. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει καν προσφορά προϊόντων για αγορά ηλεκτρονικά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο ακόμη. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα βεβαίως το ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο χρόνο χρειάζεται για να εξετάσει εντελεχώς το ζήτημα. Όμως, υπάρχουν δύο νομοθέτες. Ο δεύτερος είναι το Συμβούλιο. Και ποτέ δεν είναι καλό να βραδιπορούμε σε σύγκριση με το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντική δηλαδή και η συνεργασία μεταξύ των δύο νομοθετικών οργάνων. Αν το ένα προχωρήσει πιο γρήγορα από το άλλο, τότε αυτό μπορεί να κατοχυρώσει κάποια πράγματα αν θέλετε. Ευχαριστώ Μπάρτο. Θετική και ενθαρρυντική η παρέμβασή σας για αυτό το Magnus Opus. Θα δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Κρέσπο, για να μας πει αν μπορούμε να εναρμονίσουμε τα χρονοδιαγράμματα των δύο οργάνων. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Λοιπόν, εμείς ε, δεν θέλουμε να κάνουμε αγώνα δρόμου με το Κοινοβούλιο, με κανένα τρόπο. Θα περιοριστώ να σας δώσω τις πληροφορίες πώς έχουν οι εργασίες αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, πού βρισκόμαστε. Οι πληροφορίες που σας έδωσα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με αυτές συνήθε η ομάδα εργασίας ε, διάφορες φορές και είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τις ε, προτάσεις των κρατών μελών σε σχέση με την πλειοψηφία των κεφαλαίων της οδηγίας, με εξαίρεση το κεφάλαιο 5. Κατά την διάρκεια αυτής της ε, περίοδου είχαμε την ευκαιρία να δούμε ποιες δυσκολίες σε κάθε βήμα αντιμετωπίζαμε σε σχέση με την αρχή της ε, μέγιστη, του μέγιστου εναρμονισμού σε σχέση με τα κεφάλαια και τα κεφάλαια της πρότασης. Γνωρίζετε πολύ καλά αυτή τη δυσκολία εσείς, επειδή την αξιολογήσατε βήμα-βήμα μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Και σε εμά το ίδιο συνέβη. Τι ίδιε δυσκολίε είχαμε. Πέρα από αυτή την εργασία επί τη ουσία, σε βάθο από την Προεδρία, προσπαθήσαμε τι πέντε αισθήσει μα να τι επικεντρώσουμε στο τι γινόταν στα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών λάβαμε τη γνωμοδότηση του, της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής που ευχαριστούμε που είναι παρούσα. Σημειώσαμε τις παρεμβάσεις ε, του Ευρωβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου αυτής της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σας και της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Προσέξαμε ιδιαίτερα τις ε, τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων μερών σε όλες τις ακροάσεις που έγιναν Ακούσαμε τις απόψει των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης εδώ σε αυτή την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου και ακούσαμε με ενδιαφέρον τις τελευταίες παρεμβάσεις τη Αντιπροέδρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της κυρίας Ρέντινγκ στην έδρα της ε, ε, εδώ στις Βρυξέλλες και προβληματιστήκαμε με όλα αυτά και σκεφτήκαμε σε βάθος τα προβλήματα και αποφασίσαμε να προτείνουμε μια πολιτική συζήτηση στους Υπουργούς επικεντρωνόμενοι στο επίπεδο εναρμονισμού που θεωρούσαν οι Υπουργοί ότι ήταν αναγκαίο να επιτευχθεί σε αυτή την πρόταση. Αυτή η συζήτηση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και σε αυτή τη συζήτηση έγιναν τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, Ερωτήθηκε αν ε, η κύρια αρχή της οδηγίας θα έπρεπε να είναι η πρόταση του μέγιστου εναρμονισμού ή αν θα προτιμούσαμε μια επικέντρωση μεικτή, μια μεικτή προσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση μια πλειοψηφία των κρατών μελών ήταν υπέρ μιας ρεαλιστικής, ε, ελαστικής, μεικτής προσέγγισης και ανάλυσης ε, βήμα προς βήμα όλων των στοιχείων και κεφαλαίων της οδηγίας. Δεύτερον, ερώτημα σε σχέση με το επίπεδο εναρμονισμού που θα δίναμε στην πρόταση για το τι είδου συμβάσει θα θέλαμε. Ελάχιστο εναρμονισμό σε σχέση με τι συμβάσει που θα συνάπτονται όσον αφορά το ένα κατάστημα, εμπορικό κατάστημα και μέγιστο εναρμονισμό σε σχέση με τι συμβάσει, ε, τι εξ αποστάσεω. Η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών στο Συμβούλιο ήταν αντίθετη στο να θεσπιστούν διαφορετικά συστήματα σε σχέση με διαφορετικές συμβάσεις. Και τέλος, ερώτηση τέθηκε στους υπουργού, αν ήθελαν να εναρμονιστεί η πληροφόρηση στις τήλες συμβάσεις, στις τήλες αγορές ή αν θα έπρεπε να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ή να πηγαίνουν και πιο πέρα σε σχέση με την θέσπιση πιο αυστηρών υποχρεώσεων για την ενημέρωση και πληροφόρηση. Εδώ υπήρξε διαχωρισμό ε, διχασμός όσον αφορά τι απόψει για αυτού του είδου τι συμβάσει. Στις εβδομάδες που απομένουν ως Προεδρία για την Ισπανική Προεδρία θα συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της Βελγικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει, θα πάρει τη σκητάλη από τη δική μας Προεδρία και ο στόχος μας θα είναι να εκπονήσουμε ένα κείμενο που θα είναι παγιωμένο και ολοκληρωμένο με προτάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να σημειώσουμε πρόοδο. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Uh, well, I'd like to uh, thank you, Mr. Crespo, very much. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Κρέσπο που ήρθατε και που μας ενημερώσατε. Και ίσως και να είναι τελευταία φορά που είστε εδώ ως εκπρόσωπος της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε την, ε, με προσήλωση την εργασία σας στο Συμβούλιο. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα εγώ και οι συνάδελφοι. φαίνεται πως βρισκόμαστε σε παρόμοια σημεία εξέλιξη στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι εσείς στη Βελγική Προεδρία θα θερήσετε να συνεργαστείτε στενά με τον εισηγητή. Ανταλλαγή απόψεων που αναφέρατε ήταν δημόσια. Ε, και η γραμματεία μας που εργάζεται πολύ σκληρά έχει μάλιστα συντάξει σχετικά πρακτικά στα αγγλικά και θα τα κυκλοφορήσουμε για ενημέρωση των μελών. Δεν είναι τα ακριβή πρακτικά, απλά θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη και ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο για να δείτε και ποιες ήταν οι απόψεις των διαφόρων κατών μελών. Να το πάρετε κι εσείς. Ελπίζω πως θα συνεχίσει η Προεδρία να καλεί τον εισηγητή, γιατί έχουμε σημαντικές ιδέες για το πώς θα φτάσουμε σε κάποιες ε, ε, συμβιβαστικές, καλές συμβιβαστικές λύσεις. Να δώσω το λόγο τώρα στον Αντρέα Σβάμπ για να συνοψίσει και ίσως να σχολιάσει και το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Σβάμπ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν από πλευρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που παρόλη τη δυσμενή χρονική συγκυρία κατάφεραν να εξοικειωθούν σε αυτή την πρόταση και έδωσαν αξιόλογες προτάσεις για την περαιτέρω διαβούλευση. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Για το χρονοδιάγραμμα. Το δικό μου χρονοδιάγραμμα έχει την εξή μορφή. Στις 23 ε, Ιουνίου θα δώσω τη δεύτερη μορφή της έκθεσης που θα ολοκληρώνει την έκθεση. Τον Ιούλιο θα έχουμε αρκετό ε, χρόνο να συζητήσουμε και τα δύο τμήματα τη έκθεσής μου. Και έτσι συνολικά περίπου δύο μήνες θα έχουμε χρόνο να διατυπώσουμε τροπολογίες. Αν θέλετε για την προθεσμία τροπολογιών να είμαστε πιο ελαστικοί και να μεταθέσουμε την προθεσμία δεν έχω πρόβλημα. Αυτό που θέλω είναι στο τέλος τέλος να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Κατά, κατά αυτό λοιπόν, αυτό μπορώ να υποστηρίξω τις επιθυμίες σας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, είναι μια δουλειά που στο τέλος τέλος σε πολλές, πολλές λεπτομέρειες, σε κάποια κόμματα και κάποιες κεραίες ε, μπορεί να ε, εξαρτηθεί από κάποιες λεπτομέρειες. Μπορούν πολλά να βελτιωθούν. Όμως φυσικά έχουμε, έχουμε σκεφτεί με όριμο τρόπο αρκετά πράγματα και δεν είναι δυνατόν όλα να αλλάξουν. Ένα πράγμα είναι σαφές όμως. Δεν μπορούμε όλα να τα πετύχουμε. Δεν μπορούμε για όλες τις συμβάσεις να έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις να έχουμε ελάχιστες ρυθμίσεις ε, αλλά και να έχουμε και για όλες τις ε, συμβάσεις ε, το ίδιο πρότυπο όπως προτάθηκε από το Συμβούλιο. Αν κάποιος γνωρίζει σοβαρά την πρόταση με την οποία όλους μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε ταυτόχρονα μου δώσει αυτή τη μαγική συνταγή, αυτό το μαγικό ραβδάκι. Εγώ δεν το ξέρω ποιο είναι. Στο τέλος τέλος πρέπει να επιλέξουμε κέντρα βάρους στα οποία θα επικεντρωθούμε πιστεύω ότι αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφο Κρότσμαν, δηλαδή για τη διαφάνεια των ρυθμίσεων και των διατάξεων που θα πρέπει να αποβαίνει προ όφελο όλων. Ακόμα και αν δεν βρεθούμε στο μέγιστο επίπεδο ενό κράτου, πρέπει αυτό να είναι ο στόχο μα. Δεν είναι όμω εφικτό σε όλου του τομεί. Γι' αυτό η πρότασή μου είναι και θεωρώ ότι είναι σωστή η διαφάνεια και μπορώ νομίζω να τα επεξηγήσω και περισσότερο στην οδηγία πλαίσιο παραπάνω να έχουμε την πρόταση όπως εγώ σας την υποβάλλω σήμερα στο κεφάλαιο 2 το doorstep selling για παράδειγμα πλήρως να ενταχθούν έτσι και αυτές οι δύο οδηγίες να καταργηθούν στη συνέχεια. Απομένουν οι δύο υπόλοιπε οδηγίες για το κεφάλαιο 4 που πρέπει να ε, ε, ε, εξεταστούν και για την οδηγία για τα, τους εμπορικούς όρους των πωλήσεων στο κεφάλαιο 5. Για αυτούς τους λόγους προτείνω για πρακτικούς λόγους να πάρουμε εκείνους τους τομείς ε, όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτόν με ενιαίο τρόπο και να, τις, να κατοχυρώσουμε αυτές τις διατάξεις στην οδηγία πλαίσιο, ώστε να έχουμε για τον ελάχιστο εναρμονισμό εκείνα τα οποία θα πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τον ελάχιστο εναρμονισμό σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Δεν έχω όμω κάποιε τροπολογίε που να έχω προτείνει εγώ σχετικά. Διότι ο στόχο τη ενιαία εσωτερική αγορά θα πρέπει να είναι από τι επιθυμίε να περάσουμε στην υλοποίηση των επιθυμιών και στην πραγματοποίηση των επιθυμιών. Ακούγοντα τι συζητήσει στο Συμβούλιο και στο δημόσιο χώρο όπω έγιναν τον τελευταίο καιρό, πάντα το εξή είχαμε μπροστά μα. Αφενό, ή δυνατόν όλα να ενιοποιηθούν και να εναρμονιστούν ή να αφαιθούν όλα διαφορετικά ώστε το τέλος τέλος τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν. Αυτά όμως τα δύο δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Θα ε, ήθελα να πω ότι χαιρετίζω την προσέγγιση και θα ήθελα να πω ότι έχουμε παρόμοιες δυσκολίες και εμείς σε σχέση με τη συζήτηση όπως και το Συμβούλιο. Γι' αυτό στο πρώτο τμήμα το οποίο ολοκληρώνεται και το οποίο βασίζεται στο δικαίωμα ανάκλησης ή επαναχώρησης και στο δικαίωμα ενημέρωσης πληροφόρησης αυτά τα περιεχόμενα των δύο οδηγιών δηλαδή με αυτόν τον τρόπο μετα, ε, εδώ. Μετά περνάμε στο κεφάλαιο 5 και ασχολούμαστε με τα θέματα εκείνα που από τις υφιστάμενες οδηγίες για τα καταναλωτικά αγαθά μπορούν να ε, ρυθμιστούν. Εδώ η, η κυρία Τούν είπε ότι υπάρχει περίπλοκος χαρακτήρας επελέγησαν αυτά τα πράγματα όχι επειδή ε, είναι το χρώμα το πράσινο το θελκτικό αλλά επειδή είναι ένα θετικό μήνυμα ας το πω έτσι αυτό και θέτει το ε, σωστό βάρος. Τώρα αν ο περίπλοκος χαρακτήρας αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο ε, με τους σκιώδεις ε, εισηγητές έχω συζητήσει το θέμα, δεν θα ήθελα να διαφωνήσω. Καλύτερο θα ήταν να είχαμε μία ενιαία ρύθμιση για όλα, αλλά δεν γινότανε. Το σκέφτηκα αυτό πρόταση στην αρχή και είπα να εξετάσω όλες τις δυνατότητες εναρμονισμού και να τις εντάξω για όλους τους διαφορετικούς τομείς. Ε, τι θα γινόταν σε σχέση με το άρθρο 4. Φοβήθηκα όμως ότι η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα οδηγούσε σε κάποιες ας το πω έτσι οικοτολογίες. Ποιοι συνδυασμοί προτάσεων θα μπορούσαν να γίνουν και δεν ήθελα να επιβαρύνω τη συζήτηση. Γι' αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Ή θα αφήσουμε κάποιους τομείς ε, στο ελάχιστο, στον ελάχιστο εναρμονισμό σε σχέση με τις υφιστάμενες οδηγίες ακόμα και αν τροποποιηθούν κάποια πράγματα ή θα τις περάσουμε στην ε, ομπρέλα, στην ε, ας το πω έτσι συνολική ρύθμιση για ε, διευθέτηση. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν θα ήθελα τώρα στη συνέχεια να εξετάσω. Ένα σημείο όμως το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος Χάμπορ για τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι καταναλωτές ε, ρυθμίζουν αυτά τα θέματα σε σχέση με τις ε, πιστώσεις. Όμως, ε, όπως και αναφέρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, έχουμε και υπηρεσίες που όταν βρίσκονται κάτω από 200 ευρώ δεν ρυθμίζονται και γι' αυτό το δικαίωμα ανάκλησης ε, θα μπορούσε να εισαχθεί. Είναι σημαντικό να δει κανεί ε, το ε, σύνθετο οικοδόμημα αν σε σχέση με την οδηγία του 2000 θα μπορούσαμε να την εξετάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω τεχνικές λεπτομέρειες να μας επιβαρύνουν, αυτό μπορούμε να το κάνουμε υστερότερα. Ελπίζω ότι στις 22 Ιουνίου με το δεύτερο τμήμα, το οποίο ελπίζω ότι και νωρίτερα ακόμα θα μπορέσω να το παρουσιάσω, αλλά εξαρτάται σε κάποιο βαθμό τι θα γίνει με τις μεταφράσεις ε, και πώς θα τα καταφέρουμε. Προσπαθώ όσο το δυνατόν το γοργότερα να μπορέσω να τα υποβάλω αυτά και να λειτουργήσουν οι μεταφράσεις και χωρίς σφάλματα. Όμως ε, όλα αυτά πιέστηκαν πολύ χρονικά στο πρώτο τμήμα και υπήρξαν σφάλματα. Χαίρομαι στις κριτικές παρατηρήσεις που θα στοχεύουν προς το μέλλον και τη διευθέτηση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω για το έργο σας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να συνεργαστείτε με τη γραμματεία και τους σκιώδεις εισηγητές. Είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μία ακόμη εξωτερική διαβούλευση. Αυτό πρέπει να το αποφασίσετε εσείς. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα εργαστήριο εκτός των τακτικών συνεδριάσεων. Όσον αφορά την προθεσμία για τις 23 Ιουνίου, θα πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο στην ε, διάθεσή μας και για να εξετάσουμε τα όσα ακούσαμε σήμερα, αλλά και για την επόμενη φάση του έργου σας. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ όλους όσους ε, συνεισέφεραν σήμερα και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή. Κύριε Ζουβάν, με συγχωρείτε που πιέζω το δικό σας ε, θέμα, αλλά πρόκειται για πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Ρούλε όμως, ε, η σκληρά εργαζόμενη επί του προϋπολογισμού, θα ήθελε να μας παρουσιάσει τα πιλωτικά προγράμματα. Θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ να μην κάνετε θόρυβο όταν φεύγετε. Πολύ σύντομα, απλά για να ξέρετε πώς αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις για τον προϋπολογισμό. Έχουμε μια νέα διαδικασία μέσω της συνθήκης Λισαβόνας και μέσω της σχετικά καθυστερημένης εκλογής ε, της Επιτροπής. Και έτσι ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο κοινοβούλιο. Σε δύο φάσεις θα συζητήσουμε τα πράγματα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αφενός σήμερα έχουμε υπόψη και το συζητήσαμε με τους συντονιστέ για την Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουμε να διατυπώσουμε τροπολογίες για τα pilot projects, τα πιλωτικά προγράμματα. Θα υποβληθούν στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τα εξετάσει και θα δει πώς θα διατυπωθεί η άποψή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Pilot projects and in preparative action και ε, πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Και έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα εξέτασης και ε, ψήφισης ε, προς έγκριση. Όμως για την προπαρασκευή έχει νόημα σήμερα να αποσαφηνίσουμε αυτά τα πράγματα για τα πιλωτικά προγράμματα και να υποβάλουμε αυτές τι προτάσεις στην Επιτροπή Προπολογισμών ώστε να περάσουν μετά στην Επιτροπή. Προτείνω εξ ονόματο της Επιτροπής τρεις δράσεις να κάνουμε. Αφενός τα πιλωτικά ε, προγράμματα όπω ε, όπως τα είχαμε αποφασίσει η η κυρία Τόν ήταν αρχικά, το θυμόσαστε αυτό και υποβάλλουμε πρόταση σχετικά. Μετά έχουμε συμπληρωματική πρόταση για το θέμα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για το κείμενο Κρέξ και θέλουμε να προτείνουμε μια, ένα κονδύλιο 200.000 ευρώ για το συνολικό τομέα. Για την απογοήτευση που έχουν οι πολίτες με την ενιαία εσωτερική αγορά να γίνει από το ευρωβαρόμετρο, ε, ε, από το ευρωβαρόμετρο μια σφιγμομέτρηση, μια μελέτη πώς αντιμετωπίζουν αυτή την, απο, Πώ διαμορφώνεται η απογοήτευση των πολιτών με την ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα όμως ξεχωριστά θα το θέσουμε ως αίτημα και αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχωριστά αντίδραση γι' αυτό και μετά ακολουθούμε την ομαλή διαδικασία, την κανονική διαδικασία όπως ήδη έχει συζητηθεί για τις προ... Ε, προπαρασκευαστικές ε, δράσεις για τον τομέα, μια στιγμή να το βρω, ναι ακριβώς, για το scoreboard, τον κατάλογο επιδόσεων, τη βαθμολογία επιδόσεων. Και εδώ τώρα η η κυρία Χέτ και αυτό προτείνεται να γίνει. Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω. Αυτά θέλουμε να καταθέσουμε μέχρι τις 12 η ώρα για να τηρηθεί η προθεσμία ε, κατάθεσης των προτάσεων και μετά μπορούμε το Σεπτέμβριο τελικά να κάνουμε την ολοκληρωμένη συζήτηση. Well, I don't think we need any discussion on that, uh, really. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε. Από όσο γνωρίζω αυτές οι προτάσεις θα πάνε στην Επιτροπή. Στο φόρουμ της εσωτερικής αγοράς επανεξέταση των 20 βασικών προβλημάτων των πολιτών. Επίσης έχουμε και τον πίνακα βαθμολογίας, τον scoreboard. Χαίρομαι που έχουμε και την αρμόδια σήμερα εδώ και βεβαίως ε, θα έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε από όλων αυτών το Σεπτέμβριο. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε τώρα. Διαφωνείτε κύριε Βάλτεκα? Όχι με τις προτάσεις. Τότε δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε λέει ο Πρόεδρος. Στην ομάδα μας Συμφωνούμε με τις προτάσεις, αλλά έχουμε ένα σχόλιο για τη δεύτερη πρόταση. Εκεί που αναφέρεται ότι οι 20 βασικές πηγές ε, μη ικανοποίηση ε, των πολιτών από την εσωτερική αγορά, θα θέλαμε να προσθεθούν και οι επιχειρήσεις, ειδικά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από τους πολίτες δηλαδή. Ίσως θα έπρεπε να το συνδέσουμε αυτό γιατί νομίζω ότι αυτό δείχνει καλύτερα το τι είναι το πιλωτικό μας πρόγραμμα. Δεν ήθελα να σας χαλάσω το πρόγραμμα αλλά είναι πολιτικό. Συμφωνώ απόλυτα και θέλω να δείξουμε κατανόηση. Σχετικά γρήγορα υποβλήθηκε αυτή η πρόταση και δεν μπορέσαμε να διαβουλευτούμε επαρκώς. Αλλά είναι πολύ ευπρόσδεκτη η διόρθωση αυτή την δέχομαι ευχαρίστω και από τους κοιόδης εισηγητές των διαφορετικών ομάδων έχω την ε, είδηση ότι υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ωραία, μπορούμε να προσθέσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα το συζητήσει και η Κομισιόν μαζί μας. Υποθέτω ότι έτσι θα αναμειχθούν και οι συνάδελφοι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ επιχειρήσεων και νομίζω ότι αυτό θα είναι καλό. Τώρα, περνάμε σε ένα νέο έργο ακόμη, μία νέα έκθεση πρωτοβουλίας από τον κύριο Ζουβάν που ασχολείται με ορισμένους νέους τομείς. Έχουμε μεν κάποιους κανονισμούς για τη διαφήμιση, ειδικά όσον αφορά τις αθέμητες πρακτικές, αλλά δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ λεπτομερώς. Ο κύριος Ζουβάν είναι ο εισηγητής, ενδεχομένως ενδιαφέρεται να μας θέσει κάποιες βασικές διαστάσεις του θέματος και αν έχουμε χρόνο, ίσως οι σκιώδεις, ο κύριος Στανζάρη είναι εδώ, ο κύριος Ροσφόρ είναι. Από τους πράσινους δεν ξέρω ποιος θα είναι ο σκιώδης, ο κύριος Κιγιόν δεν είναι εδώ, ίσως μπορεί να τον αντικαταστήσει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Από τους πρασίνους και τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα είναι ο σκιώδης. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ζουβάν, μπορείτε να παρουσιάσετε την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τίτλος είναι «Συνέπειες ε, της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών». Ξεκινάω με λίγα λόγια για τη μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να παρουσιάσουμε την έκθεση στην ε, ΙΜΚΟ τον Ιούλιο, μάλλον 12 Ιουλίου. Προθεσμία για τις ε, τροπολογίες στην ΙΜΚΟ αρχές ε, Σεπτεμβρίου, ώστε να περάσει από την Ολομέλεια Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών ενώ έχουμε ζητήσει και σημειώματα επεξηγηματικά από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για την οδηγία για τις ε, αθέμητες ε, διαφημιστικές πρακτικές αλλά και για τις ε, πολύ μέσω διαδικτύου και περιμένουμε αυτά τα σημειώματα αρχές Ιουλίου. Επί της ουσίας τώρα. Πρόκειται για περίπλοκο και πολύ ευρύ θέμα. Είχαμε μία συνεδρίαση με τους Κιώδης την προηγούμενη εβδομάδα. Να πω καταρχάς ότι πρέπει να δούμε και τα θετικά και τα αρνητικά της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών, γιατί δεν είναι μόνο αρνητικός ο ρόλος τα θετικά πέρα από το ότι διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα η διαφήμιση και αυξάνει τον ανταγωνισμό, επιτρέπει τη μείωση των δεσπόζουσα της δεσπόζουσας δίνει επιλογές στους καταναλωτές από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες. Έχουμε βεβαίως ε, τις ε, υπερβολικές διαφημίσεις, τις διαφημίσεις που ψεύδονται κτλ. Υπάρχει και θέμα μόλυνσης αν θέλετε και του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο του πολίτη η λήψη spam, email λοιπά, η διαφήμιση από τη μία πλευρά μπορεί να αποφύγει τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης, από την άλλη όμως όταν μία εταιρεία θέλει να μπει στην αγορά είναι υπερβολικές και πολύ ψηλές οι διαφημιστικές δαπάνες που απαιτούνται. Άλλο θέμα είναι οι ευάλωτοι στόχοι. Παιδιά, για παράδειγμα, μια κατηγορία του πληθυσμού που μπορεί να υποφέρει ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες της διαφήμισης. Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά τις αλλαγές στα ΜΜΕ. Οι νέες τεχνολογίες ενημέρωσης, οι νέοι τρόποι διαφήμισης, τους οποίους δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε πριν από κάποια χρόνια, παίζουν πολύ μεγάλη ρόλο. Για παράδειγμα, έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, που επιτρέπουν τη διαφήμιση να εισδύσει στον ιδιωτικό μας κόσμο, στην ιδιωτική μας σφαίρα, με έναν τρόπο που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν. Οι εταιρείε ανοίγουν ένα προφίλ στο Facebook και έχουν πλέον ε, πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο ατόμων. Και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ρύθμιση εκεί. Αύριο που θα έχουμε και άλλους τρόπους και που θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω τηλεόρασης, τηλεφώνου κτλ. Θα έχουμε και επίσης τη διασύνδεση της τηλεόρασης και του διαδικτύου και αυτό σημαίνει ότι αν εσείς έχετε γράψει τα γούστα σας, έχουν δει τα γούστα σας από το διαδίκτυο, θα λαμβάνετε στην τηλεόρασή σας στοχευμένες διαφημίσεις. Θα μπορούν να ψάξουν τις λέξεις κλειδιά που έχετε ψάξει στο ίντερνετ ή ακόμη και σε μία τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχατε για να λάβετε διαφημίσεις για άλλα θέματα. Έτσι αν είχατε παραγγείλει μία πίτσα από το τηλέφωνο θα μπορούσατε να λάβετε σχετικές διαφημίσεις. Βλέπουμε ότι σήμερα το Google και άλλες εταιρείες αναλύουν τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε αναζητήσεις, για να μας στέλνουν στοχευμένες διαφημίσεις. Πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο και να θέσουμε και ερωτήματα που δεν είχαν θεθεί στο παρελθόν. Είναι αλήθεια ότι είχαμε ασχοληθεί και είχαμε επιλύσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν, για παράδειγμα με την οδηγία για τις αθέμητες πρακτικές. Όμως τώρα έχουμε και νέα ερωτήματα που τίθενται και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κείμενο και για να τονίσουμε τα όσα ήδη ισχύουν, για παράδειγμα όσον αφορά την επιθετική διαφήμιση, την ψευδή διαφήμιση, να εξετάσουμε δηλαδή κατά πόσο είναι κατάλληλα τα εργαλεία που ήδη έχουμε, πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της αυτορύθμισης, που είναι ενδιαφέρουσα λύση, αλλά είναι πολύ ετερογενής αυτή τη στιγμή. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για πολύ πολύπλοκο θέμα και συνεχώς μεταλλασσόμενο. Δεν είναι ομοιογενές. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε ερωτήματα που δεν είχαν τεθεί στο παρελθόν, ακόμη και αν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη τεχνική λύση να προτείνουμε. Για παράδειγμα, οι κρυμμένες διαφήμισης στο διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα που συζήτησα με Δεν έχουν ακόμη λύση οι εμπειρογνώμονες. Όμως υπάρχει αυτή η πρακτική. Έχουμε εταιρείες που ενδεχομένως ε, τους που ενδεχομένως οδήγησαν κάποιους καταναλωτές να κάνουν αρνητικές κρίσεις, ενδεχομένως άθελά τους για κάποια προϊόντα και που αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για διαφήμιση. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα θέματα που με απασχολούν στην έκθεση και ανυπομονώ να έχω καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους χειώδεις συζητητές. Συμφωνούμε μαζί σα ε, να έχουμε μια επικεντρωμένη, στόχοθετημένη έκθεση και κάποια από τα θέματα που αναφέρατε ήταν πολύ θελκτικά. Και επίσης ε, θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Θα έχει ευρύτερη επίπτωση σε πολλές γενικέ διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπής που συσχετίζονται σε σχέση με την κοινωνία της αγοράς. Χαίρομαι ιδιαίτερα να έχουμε τον τον κύριο εδώ που θα μπορέσει να μας πει δύο λόγια. Τον καλωσορίζω. Ανάμεσά μας έχουμε χρόνο νομίζω για μια πρώτη επαφή σκιωδών εισηγητών που θα αντιδράσουν σε αυτές η κυρία Γκέπαρντ, ο κύριος Χοσφό, η κυρία Ρούιλε μετά και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, η ε, κυρία Γκέπαρντ πρώτη λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε δυστυχώς παρακολείται ο σκιώδης εισηγητής μας ότι πρέπει να είναι σε άλλη συνεδρίαση και ζητεί συγγνώμη για το ότι δεν μπορεί να παραστεί και συζητήσεις και τα λοιπά κάποια μου έχει δώσει να πω κάποια στοιχεία που θα μπορούσα να αναφέρω. Δεν τα χρειάζομαι όμως αυτά, επειδή όλα αυτά έχουν ήδη αναφερθεί και γι' αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς αυτά τα κέντρα βάρους τα οποία προαναφέρατε και η νέα ε, δυνατότητα επικοινωνία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι οι απαντήσεις που θα δώσουμε. Δεν πρόκειται μόνο σε σχέση με το διαδίκτυο, αλλά πρόκειται και για αυτές τις σελίδες που ε, πάντα βρίσκονται μπροστά μας όταν θέλει κανείς να δει κάποια πράγματα. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν που πρέπει να ρυθμιστούν. Αναφέρατε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή πολύ λίγο συζητείται, που όμως πιθανότατα όλο και περισσότερο θα διαδραματίζει ένα ρόλο. Και αυτό είναι αυτές οι σελίδες που προσφέρονται και που παρουσιάζονται και είναι συγκαλυμμένες διαφημίσεις και κανείς δεν μπορεί να δει άμεσα ότι είναι διαφημίσεις. Εμφανίζονται σαν κάτι πιο σοβαρό, σαν ενημέρωση, πληροφόρηση των πολιτών. Και αυτή τη συζήτηση την είχαμε και πρόσφατα και σε σχέση και με τα ιατρικά προϊόντα, τα σκευάσματα, τα φάρμακα στο διαδίκτυο και τέτοιου είδους ε, συγκαλυμμένη διαφήμιση και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υφέρπουσας ή ε, συγκαλυμμένης διαφήμισης στο διαδίκτυο που δεν δίνει πραγματικές πληροφορίες αλλά είναι απλά διαφήμιση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κάποια πράγματα να γίνουν και κάτι να κάνουμε. Επίσης αναφέρατε θέματα που συσχετίζουν με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Συγγνώμη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί σε αυτόν τον ψηφιακά παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς και πιο έντονα ασχολείται και θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Στη συνέχεια με την κυρία Κρός θα συζητήσουμε, αλλά και η κυρία Ρέντινγκ εχθές στην, ε, στο φόρουμ στην ημερίδα προστασίας των καταναλωτών το είπε με κάθε σαφήνεια κάθετα, ότι αυτό θα είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα την απασχολήσει και θέλει να το ρυθμίσει τι θα κάνουμε σε σχέση με αυτό. Και θα έλεγα λοιπόν ότι ε, στις παρουσιάσεις που δώσατε εσείς πραγματικά μια πολύ καλή εικόνα, παρουσίαση δόθηκε. Και θα έλεγα ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε. Ευχαριστώ. Uh, ε, Mr. Ο κύριος Ροσφόρ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό την πολύ ταχύ εξέλιξη. Η παρουσίαση του συναδέλφου Ζουβέ ήταν εξαιρετική και φυσικά δεν είμαστε κατά, δεν είναι κανείς κατά της διαφήμισης. Ίσως ε, να αποτελεί ένα εργαλείο δημιουργικότητας ε, μεγάλες σύγχρονες επιχειρήσεις και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Να, ήθελα απλά να πω ότι υπάρχουν δύο παρατηρήσεις που είναι πολύ σημαντικές. Η μία είναι αυτή που αναφέρθηκε. Είναι, σύντομα είναι ότι συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Ζουβάν και η κυρία Κέπχαρτ, αλλά εσείς επιφέρετε μια πολύ μεγάλη καινοτομία Μέχρι στιγμή αυτό που κάνουν οι επιχειρήσεις και πολλοί πάρα πολύ το κάνουν υπό τη μορφή διάδοση πληροφοριών μέσω των δικτύων και μέσω του Ιντερνετ δεν θεωρείται διαφήμιση. Αν λοιπόν στο τέλος των εργασιών καταλήξουμε και πούμε ότι αυτό εμπίπτει στο πεδίο της διαφήμισης θα ήταν μια αλλαγή στον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Για να είμαστε ξεκάθαροι, οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα σε αυτό που ονομάζουν υπηρεσία εξωτικής επικοινωνίας έχουν διάφορους που αποτελούν το, ένα είδος ε, φρουρού και που στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και δεν είναι στον ίδιο τομέα, δεν είναι στην ίδια υπηρεσία της διαφήμισης ή των δημοσίων σχέσεων. Θα πρέπει λοιπόν να, να καταλάβουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το business, το business της ε, διαφήμισης με την παραδοσιακή του έννοια. Να πούμε ότι αυτές που είναι οι δαπάνες εκτός ΜΜΕ είναι πιο σημαντικές από αυτές που είναι εντός. Το mailing και το e-mailing και τα λοιπά ήδη ε, για τις επιχειρήσεις είναι πιο σημαντικό στο μέσο δαπανών από ότι οι παραδοσιακές διαφημίσεις. Και κάτι ακόμα που θέλω να αναφέρω και το είπε ο κ. Ζουβά Μιλάμε για το αν η αυτορύθμιση αρκεί ή αν πρέπει να υπάρχει δημόσια ρύθμιση. Το έχουμε αυτό, το συζητάμε με τις, ε, ε, τους οργανισμούς ε, πιστοληπτικής αξιοπιστίας ε, και διάφορα άλλα. Μιλάμε για τους ε, επίση υπάρχουν οι επαγγελματίες που στην ουσία δημιουργούν ένα είδος αστυνομίας, αστυνόμευσης του επαγγέλματό τους και άρα θα πρέπει να διερωτηθούμε αν η αυτορύθμιση αρκή ή όχι. Ίσως θα ξέρετε ότι είναι μανία μου αυτό και ιδιαίτερα προσφυλές μου θέμα, ότι δεν είναι, υπάρχει μόνο το θέμα της επαιδείας ε, του και της ενημέρωσης καταναλωτή και στο θέμα της διαφήμισης είναι πολύ σημαντικό και η υπόθεση. Σε οποιαδήποτε ομάδα ε, μαθητών 13 με 14 χρονών πάντα λέω πώς να αποκοποδικοποιούν την διαφήμιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κατά της διαφήμισης, απλώς σημαίνει ότι έχουμε μια σχέση ευφυή με τη διαφήμιση και μας επιτρέπει αυτό αργότερα να μπορούμε να καταναλώνουμε έχοντας έχοντας γνώση του θέματος. Ευχαριστώ. Πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες ήδη ακούγονται. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Η κυρία Ρούλε, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλω μια πρόσθετη ιδέα να δώσω. Αφενός θεωρώ πως και ο κύριος Ροσφόρ ότι θα έπρεπε να δούμε ότι υπάρχουν σημαντικές μεταθέσεις οικονομικών ροών εδώ και η χρηματοδότηση για παράδειγμα των παραδοσιακών μέσων και των ραδιοφωνικών μέσων πιέζονται, τίθενται υπό ιδιαίτερη πίεση τα παραδοσιακά μέσα και πρέπει να δούμε και τα θέματα χρηματοδότησης και αυτό διαδραματίζει ένα ρόλο που πρέπει να εξετάσουμε αλλά και τα δικά μας μέσα και εργαλεία πρέπει να εξετάσουμε παράδειγμα και αυτό το κοινοβούλιο και άλλα κοινοβούλια προσπαθούν όλο και περισσότερο στις διαφημίσεις τις πληροφορίες να τις κατοχυρώνουν σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο να προβλέπεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά πληροφορίες ξεχωριστά από, την, από τη διαφήμιση. Έχουν υπόψη όμως την παραδοσιακή διαφήμιση. Εδώ να επιβαρύνεται η διαφήμιση με επιπλέον ε, υποχρεώσεις ε, ρυθμιστικές ε, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι και τίποτα δεν ρυθμίζεται, τίποτα δεν καθοδηγούμε, όλα γίνονται χωρίς τη δική μας επιρροή. Και αυτό πρέπει κατεπηγόντως να το συζητήσουμε, γιατί εμείς ως ρυθμιστές εδώ πρέπει να δούμε ότι αλλάζει η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και ότι έχουμε πρόσθετες μεταθέσεις και αλλαγές και πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούλη, κυρία Μακλάκη. να σας πω ότι η διαφήμιση μπορεί να λειτουργήσει ως ενημερωτικό εργαλείο για τον καταναλωτή, καθώς και ε, προώθηση για τις επιχειρήσεις. Και φτάνουμε σε αυτήν την ισορροπία που είναι θέμα κλειδί. Φυσικά θα πρέπει να μεριμνήσουμε για όλες τις μορφές διαφήμισης για τα παιδιά. Ε, αλλά την άλλη θα πρέπει να προσέξουμε, είναι μια μεγάλη όθηση η διαφήμιση για τις επιχειρήσεις, για τις, ε, τα κανάλια, για τον έντυπο τύπο και για τον αθλητισμό μπορεί να έχουν δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια θετική πτυχή στη διαφήμιση, αλλά πρέπει να είναι σαφή ε, να μην είναι παραπλανητική, είτε να μην δει. Θα λέει, θα πρέπει να λέει, να κάνει αυτό που λέει στην συσκευασία. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά εργασία. και ε, πρέπει να προωθήσουμε αυτή την αγορά. Και η κυρία Σαλ Ντεμόζε. Α, συγγνώμη, ο κύριος Τρενταφυλλίδης πρώτα. Και μετά, αν θέλει ο κύριος Βερμόντι να κάνει μια σύντομη παρέμβαση και να κλείσουμε στην ώρα μας, μόλις πριν έρθει η κυρία Κρούζ. Πρόεδρε. όπως είπατε, ο κύριο Ντεγιόνγκ που είναι σκιώδης, δεν είναι εδώ, αλλά έχω ακούσει τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον εισηγητή και από τους άλλους συναδέλφου, που φαίνεται πως η συζήτηση θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο μέλλον. Φυσικά η διαφήμιση βρίσκεται στο, επίκεντρο, στο κέντρο της ζωής μας. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί σωστά. Θα το συζητήσω και με τον κύριο Ντεγιόγκ που είναι ο εισηγητής μας και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάλτε Μόζε. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να πω ότι είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τους πολίτες μας και είναι δίκαιο ε, και είναι μεγάλη, πολύ σπουδαίος κλάδος, πολύ μεγάλε επιχειρήσει, αλλά στο τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές είναι αυτοί που πληρώνουν ε, την ε, νύφη. Δεν είμαστε κατά τη διαφήμιση φυσικά, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το κόστος ε, να μην υπόγειται τη διαφήμιση χωρίς να το ε, επιθυμούν. Δεν θέλουμε ε, λοιπόν να είναι ανεξέλεγκτες οι διαφημίσεις, να, μην, να μπορεί ένας καταναλωτής που δεν το επιθυμεί να μην βλέπει τη διαφήμιση. Ε, εγώ πιστεύω πως αυτό που λειτουργεί είναι η συνρύθμιση, δηλαδή η ρύθμιση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις αρχές ώστε να φτάσουμε σε καλύτερους κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Φαντάζομαι πως θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η διαδικασία. Τζουζέπε Εβερμόντι, θέλετε να παρέμβετε από την προπτική ε, αυτού που θα λάβει πιθανότατα την έκθεση και θα πρέπει να ενεργήσει από αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουβάν που έθιξε αυτό, κύριε Ζουβάν που έθιξε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τι επιπτώσει όσον αφορά διαφημίσει στου καταναλωτές είναι κάτι που αναπόφευκτα θα πρέπει να οδηγήσει στο να δούμε όλο τον περίγυρο που αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι σε σχέση με την εφαρμογή της ε, οδηγίας ε, που πρέπει η έκθεση να υποβληθεί του χρόνου. Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση λόγω της καθυστερημένης εφαρμογής οδηγίας από τα κρατη Όμως η δική σας, ε, ο δικός σας προβληματισμός θα βασιστεί στις κατευθυντήριες γραμμές και στις ε, ε, συστάσεις ε, που βρίσκονται ήδη στη διάθεσή σας στο διαδίκτυο και που θα πρέπει να επικαιροποιηθούν υπό το φως των δικών σας διακριβώσεων και συμπερασμάτων. Βέβαια θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Δύο παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη παρατηρήση σε σχέση με την αντίδρασή μου προς τις παρατηρήσεις του κυρίου Ροσφόρ για το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο, οριζόντιο ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στις διαφημίσεις. Αφορά και εφαρμόζεται σε σχέση με όλες τις εμπορικές πρακτικές. Θεωρητικά εφαρμόζεται λοιπόν νομικά και σε εμπορικές ε, γνωστοποιήσεις ή στοιχεία ή οποιασδήποτε εμπορικές πρακτικές ε, ε, όσον αφορά το διαδίκτυο. Σίγουρα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις συγκαλυμμένης διαφήμισης ή σε ας το πω έτσι κείμενα τα οποία πληρώνονται αγοράζονται από τους διαφημιστές, πληρώνονται από αυτούς ώστε να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να περάσουν τις, ε, τα μηνύματά τους. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε μαύρο πίνακα όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές και που κατηγορηματικά και κάθετα απαγορεύεται πανευρωπαϊκά. Γνωρίζουμε βέβαια ότι καμιά φορά το ότι δεν υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό κενό, όμως ε, η κανονισμοί, κανόνες και διατάξεις θα μπορούσαν να διατυπώνονται με σαφέστερο τρόπο, με εύληπτο τρόπο, ώστε να ε, μπορούν να ε, εφαρμόζονται. Και αυτό μπορεί ιδιαίτερα να γίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Θεωρούμε ότι τα δικά σας συμπεράσματα, κύριε Ζουβά θα είναι θεμελιώδους σημασία για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κάτι άλλο τώρα το οποίο πρέπει πάντα να θυμόμαστε. Το πρώτο τελευταίο σημείο είναι αυτό και αυτό είναι το ότι μπορεί να υπάρχουν ρυθμιστικά προβλήματα. Ίσως οι κανόνες μπορεί να είναι πιο σαφείς, όμως είναι θέμα επιβολής των κανόνων κυρίαρχα σε πρώτο λόγο. Είναι ένα θέμα επιβολής, ας το πω έτσι, των διατάξεων που πρέπει να ισχύει σε σχέση με το δίκτυο των αρμόδιων του δικτύου προστασίας των καταναλωτών που πρέπει να είναι αρμόδιο και είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών διασυνοριακά, πανευρωπαϊκά. Και τέλος, ναι, το θέμα της ε, συμπεριφοράς, ε, του πώς η συμπεριφορά μπορεί να επηρεάζεται από στοχοθετημένη διαφήμιση. Αυτό είναι ένα ε, θέμα πρωτοβουλία, έκθεσης της Επιτροπής όπου θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε και στην αναθεώρηση των αθέμι, της, οδηγία, της οδηγίας περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών και την αναθεώρησή της. Θα το εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βερμόντι. Να καλωσορίσω την Επίτροπο Κρούζ. Να σας πω, Επίτροπε, ότι μιλάμε για μια νέα έκθεση που αφορά τον αντίκτυπο της διαφήμισης στην συμπεριφορά του καταναλωτή και μιλάμε και για τις διαφημίσεις online. Ξέρω ότι στο πρόγραμμα δράσης στο ψηφιακό μας έχετε μιλήσει και θα εξετάσετε κάποια θέματα για τα προσωπικά δεδομένα και την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων για την προστασία αυτών. Ε, με τα χαράς λοιπόν καλωσορίζουμε και πάλι τον Τζουζέπε Βερμόντι, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Κύριε Ζουβέ, θέλετε να κάνετε κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις. Ήδη μας εκθέσατε το χρονοδιάγραμμά σας. Για να ανακεφαλαιώσω μόνο, η προθεσμία για την έκθεσή σας για τη μετάφραση είναι η 24η Ιουνίου, εξέταση του σχεδίου έκθεσης 12 και 13 Ιουλίου, ίσως με κάποιο ενημερωτικό σημείωμα. Η υποβολή τροπολογιών είναι 11-12 Σεπτεμβρίου, ψήφος 29 Σεπτεμβρίου και στόχος είναι να εξεταστεί από την Ολομέλη στη 2η του Οκτωβρίου στην 1η του Νοεμβρίου. Αυτό συμβαδίζει και με τα όσα έλεγε ο κύριος Εβερμόντι νομίζω για την οδηγία. Θέλετε να κάνετε κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις κύριε Ζουβά. Όχι πρόεδρε, δεν μένει τίποτα άλλο παρά να στρωθώ στη δουλειά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους όσους συνέβαλαν στην συζήτηση. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ιδιαίτερη χαρά ε, που καλωσορίζουμε σήμερα την Επίτροπο Κρούς, που είναι Επίτροπος για την ψηφιακή ατζέντα για πρώτη φορά. Ξέρω πως ε, τα θέματα του καταναλωτή και της ε, εσωτερικής αγοράς είναι και τμήμα του χαρτοφυλακίου σας και Έχετε πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη εργασία για το μέλλον. Έχουμε δει και έχουμε δώσει κάποια αντίγραφα στους συναδέλφους ε, για την, ε, από το πρόγραμμά σας. Είστε εδώ για να μας μιλήσετε για το άμεσο μέλλον και το πρόγραμμα εργασίας σας. Αλλά ίσως οι συνάδελφοι να σας ρωτήσουν γι' αυτό αλλά και για κάποιες άλλες πτυχές της ψηφιακής ατζέντα επίσης. Ε, γιατί βέβαια Μέσω του προγραμματός σας θα ξεκινήσετε τα πρώτα στοιχεία για την ψηφιακή ατζέντα και θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, καθώς εξετάζουμε τις, ε, το πρόγραμμα εργασίας. Σας δίνω με τα χαρά στο λόγο και μετά θα έχουμε έναν γύρο ερωτήσεων και θα έχουμε γενικά μία ώρα στη διάθεσή μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη κύριοι Ευρωβουλευτές, κατά τα τέλη αυτής της συνεδρίασης ειλικρινά ελπίζω ότι σίγουρα θα εξακολουθείτε να είσαστε βουλευτές, ευρωβουλευτές, αλλά αντί να λέω εξοχότατοι ευρωβουλευτές, θα είμαστε πια φιλαράκια και θα έχουμε εξοικειωθεί περισσότερο. Και έτσι θα μπορέσουμε με μια εταιρική σχέση φιλική, ας το πω έτσι, σε μια φιλική ε, διάσταση συσχετισμού να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας, που έχουν τεράστια σημασία για το μέλλον. Να χαράξουμε την πορεία προς το μέλλον με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Για τους πρώτους τρίτους μήνες ε, σε αυτό το αξίωμα μπορώ να σας διασφαλίσω ότι έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί κανείς να πετύχει ως χαρτοφυλάκιο. Είναι δημιουργικό, είναι ε, οριζόντιο, εγκάρσιου χαρακτήρα, είναι εξυγχρονιστικό, συνδέεται με όλες τις δράσεις ε, στην ευρωπαϊκή μας κοινότητα και είναι ένα χαρτοφυλάκιο όπου πρέπει και χρειάζεται κανείς να συνοδεύεται στις ε, δράσεις του από πολλούς που θα υποστηρίζουν και παράλληλα θα δρουν για να στεφθεί το εγχείρημα με επιτυχία. Τούτου λεχθέντος φυσικά πραγματικά όχι μόνο ελπίζω αλλά και επιθυμώ και θα ήθελα να μπορέσετε να προσθέσετε και εσείς ε, την προσπάθεια και παρουσία σα στην προσπάθεια να καταφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Τούτου λεχθέντος κάνουμε λόγο για αυτήν την ψηφιακή ατζέντα. Εν παρόδο είναι ένα προϊόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν χρειάζεται να το επεξηγήσω σε εσά, σε άλλους όμως στους οποίους ομιλώ, πρέπει να το αναφέρω ότι δεν είναι προϊόν ενός επιτρόπου, είναι προϊόν της Ευρωπαϊκή Επιτροπής συλλογικά. Πρέπει να υιοθετώ αυτή τη γραμμή, διαφορετικά δεν θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Στο τέλος τέλος όλοι οι συναδελφοί μου επίτροποι εμπλέκονται σε αυτές τις συζητήσεις και έχοντας αναφέρει αυτό δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζομαι και την υποστήριξη της Ευρωβουλής και γι' αυτό με ιδιαίτερη χαρά είμαι εδώ ανάμεσά σας και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, όχι μόνο για το ότι μου δίνετε ευκαιρία να εξηγήσω όλα αυτά σε εσά, αλλά να έχουμε και ένα διάλογο μαζί σας και να ακούσω τις δικές σας απόψεις και τα δικά σας θέματα και ενδιαφέροντα. Και εν παρόδο δεν είναι το ε, και είναι το, ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω και το Συμβούλιο επίσης είναι σημαντικό τα Συμβούλια τα Ευρωπαϊκά, το και τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και το Συμβούλιο έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να είναι ένας συνδυασμός λοιπόν, μια συνδυασμένη δράση που πρέπει να πετύχουμε. Κατά τούτο λοιπόν από, σε σχέση με τα Συμβούλια έχουν επεξηγηθεί οι προτάσεις περί τίνος πρόκειται και υπάρχει ενθουσιασμός, ενθουσιώδης υποστήριξη. Μέχρι σε εδώ όλα καλά λοιπόν. Ας κάνουμε την ευχή και ας κρατάμε σταυρωμένα τα δάχτυλά μας να πάνε όλα καλά. Τώρα, αναφέροντας ότι είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η πρώτη ναυαρχίδα, στην την αποκαλέσουμε έτσι, αυτή της ε, πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο το φθινόπωρο ε, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Είναι η ναυαρχίδα η οποία καθελκύεται πρώτη και ξεκινά το ταξίδι πρώτη. Δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσα ναυαρχίδα, αλλά και πολύ σημαντική ναυαρχίδα αυτό το εγχείρημα και τώρα σε σχέση με όλα αυτά να πω και ένα άλλο θέμα. Τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες ή άλλα θέματα. Φυσικά μπορεί να συζητήσει κανείς και άλλα θέματα. Αλλά αυτό ήταν μία από τις γραμμές που είχα υιοθετήσει. Ας είναι σαφής η γλώσσα μας. Ας είμαστε ξεκάθαροι και ρεαλιστικοί. Όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό. Και να μην έχουμε ένα ευχολόγιο εν είδη τηλεφωνικού καταλόγου, σαν ένα τηλεφωνικό κατάλογο ε, ευρύτε, ευρύτερες δηλαδή επιθυμίες και λεπτομέρειες, αλλά ας επικεντρωθούμε στο να περάσει το μήνυμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεύτερο πρόβλημα και δυνατότητες επίλυσης ψηφιακή αγορά και η απουσία της, οι ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν ε, σε σχέση με τα δίκτυα προβλήματα, υπάρχουν ε, ελλείψεις στις επενδύσεις, υπάρχει μη επαρκής έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχει εδώ έλλειψη σε, ε, όσον αφορά την εξοικείωση των πολιτών μας με το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ψηφιακά θέματα. Πολλά πρέπει να γίνουν λοιπόν. Αν επιτρέπετε ας τα δούμε ένα-ένα. Ένα, πρώτο, κάνοντας λόγο για την ενιαία εσωτερική αγορά στα ψηφιακά όπου ψηφιακά εμπορεύματα, αγαθά, ψηφιακές υπηρεσίες θα μπορούν να είναι προσπελάσιμες και ανοιχτές σε όλους τους πολίτες, παντού. Και εδώ πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τέλη του έτους θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις, παράδειγμα, και γνωρίζω το θέμα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα συναφή. Και κάνουμε λόγο για την αγορά online, τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές με τους εμπλεκόμενους και θα υπάρξει feedback και θα υπάρξουν προτάσεις που θα εξεταστούν για αυτές όλες τις πρωτοβουλίες. Μετά, έχουμε την διεύρυνση και επέκταση του φάσματος της οδηγίας επιτρέψτε μου να μην κάνω τόσο μεγάλο άλμα και να πω πιο συγκεκριμένα κάτι άλλο. Κάνοντας λόγο για την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στόχος μας είναι να δώσουμε input για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προσοχή που αξίζει σε αυτό. Ιδιαίτερα η έκθεση του Παύλο Άριας για αυτό το θέμα. Τη συζητήσατε χθε, έτσι, έχω ενημερωθεί σχετικά. Ναι, έχω καλά ενημερωθεί από ό,τι βλέπετε. Για να καταφέρουμε μια σωστή ενιαία εσωτερική αγορά στα ψηφιακά, πρέπει να ανοίξουμε την πρόσβαση, την προσπελασιμότητα στο περιεχόμενο, στην ουσία, content. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να ε, υπάρξει η δυνατότητα δημιουργικότητας στο διαδίκτυο και ψηφιακά και προώθηση της προσπελασιμότητα στο διαδίκτυο όλων των μορφών περιεχομένου content στου χρήστε. και πρέπει να είναι θελκτική κο αυτό το πλαίσιο σε προσιτές τιμές που θα διασφαλίζει επίσης και την προστασία και την σωστή ανταμοιβή των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Είναι σημαντικό και αυτό και πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά, στον πυρήνα των συζητήσεων. Ακολουθώντας μια δημόσια ακρόαση τον Απρίλιο, ξεκίνησε ήδη τη δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια οδηγία πλαίσιο που θα διευκολύνει την ρύθμιση των θεμάτων copyright και ε, των αδειοδοτήσεων διασυνοριακά. Και θα δούμε όλες τις δυνατές ε, εφικτές λύσεις που θα μπορούν να είναι διαθέσιμες. Επίσης θα υποβάλουμε, όπως αναφέρεται στην ψηφιακή ατζέντα, στο ε, ψηφιακό θεματολόγιο, κατά τα τέλη του 2010, με μια πράσινη βίβλο που θα αναφέρει τις διάφορε δυνατότητε δυνατότητες και πρωτοβουλίες όσον αφορά τα ψηφιακά θέματα στο οπτικοακουστικό επίπεδο και τις δυνατότητες που θα έχουμε. Μέχρι το 2012 θα ξαναδούμε και θα αναθεωρήσουμε τα πράγματα, να δούμε αν περαιτέρω μέτρα θα είναι αναγκαία. Μπορείτε να δείτε εδώ λοιπόν, συνεργασία, σε συνεργασία εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς ως αρμόδιοι, σε συνεργασία με άλλους, μπορούμε να υποβάλουμε αυτές τις προτάσεις. Εμείς δίνουμε σαφή ευκαιρία και προτεραιότητα. Αν δεν λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά ή αν δεν πάνε καλά, αμέσως θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε μέσο και εργαλείο που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα πράγματα ώστε να είμαστε οι καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει και οι δύο και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, η διασφάλιση μιας ενιαίας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς σε διασυνοριακό πλαίσιο πρέπει να οδηγήσει στην ολοκλήρωση και του φυσικά ενιαίου χώρου πληρωμών. Και μια αναθεώρηση και επέκταση της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές για να υπάρχει μια δυνατότητα διαλυτικής λειτουργικότητας και αμοιβαίας αναγνώρισης ηλεκτρονικής ταυτότητας και ηλεκτρονικής υπογραφής. Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στον ψηφιακό τομέα στους πολίτες μας. Είναι κάτι όπου πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνειδητοί και ενεργοί. Δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη. Πρέπει να ξαναδούμε τα στοιχεία Προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και να θεσπίσουμε ένα διοντολογικό κώδικα μέχρι το 2012 όπου θα συνοψίζονται τα δικαιώματα των χρηστών του ψηφιακού κόσμου μέσα σε αυτό το πλαίσιο για αγορές και συναλλαγές. Επιπλέον θα ενισχύσουμε τις ε, ε, ανακοινώσεις και για τις υπηρεσίες στην, στην ε, ψηφιακή αγορά και μέσω SWIFT. Δεύτερον, η διαλειτουργικότητα και οι προδιαγραφές. Υπάρχουν ακόμα δυναμίες όσον αφορά την θέσπιση ε, διατάξεων και προδιαγραφών υπάρχουν ακόμα και αδυναμίες στις δημόσιες προμήθειες και αγορές και στο συντονισμό των δημοσίων αρχών. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερες προδιαγραφές ICT πανευρωπαϊκά. Και έτσι θα πρέπει να δούμε και την τυποποίηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο που πρέπει να προαχθεί όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και το ICT πλαίσιο για να δοθεί η δυνατότητα χρήσης από τα παγκόσμια φόρα των προδιαγραφών αυτών του ICT. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2010 θα υιοθετήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαλειτουργικότητα και ένα πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Επ' αυτόν πρέπει να βελτιώσουμε οπωσδήποτε το δυναμικό να προβλέπουμε, να δρούμε προληπτικά, να εντοπίζουμε και να αντιδρούμε έγκαιρα θέματα ασφάλειας ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει γοργά να δρούμε, πρέπει να αξιολογούμε τα μέσα μας και πρέπει να έχουμε επιμερισμένη κοινή αρμοδιότητα μεταξύ ατόμων εταιριών και ιδιωτών και στο, ε, στις χώρες μας ε, και παγκόσμια, παγκοσμιοποιημένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο θα υποβάλει μια πρόταση <clears throat> για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο όσον αφορά την, την πληροφόρηση και ασφάλεια και την ε, υπηρεσία που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων ασφάλειας όσον αφορά αυτά τα δίκτυα. Και επιπλέον θα έχουμε μια αναθεώρηση της οδηγίας ε, για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε την επίπτωση των νέων τεχνολογιών όσον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας και τον ιδιωτικό τομέα και τα ιδιωτικά δεδομένα και θα πρέπει να διαμορφώσουμε ε, τις πολιτικές μας ε, που θα πρέπει να είναι ευρύτερες. Διαφάνεια λοιπόν δίκαιος χαρακτήρας και χρήση, έλεγχος θα πρέπει να είναι οι αρχές που θα διέπουν όλους τους εμπλεκόμενους. Και φυσικά ενθαρρύνω και τις βιομηχανίες και τους ε, όσους εμπλέκονται να είναι φιλικοί προς τους χρήστες και να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές πρέπει να ολοκληρώσουν αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο με τις αντίστοιχε ρυθμίσεις. Τώρα, έχουμε και την ανάγκη γοργά, γοργής επικοινωνίας και πρόσβασης και υπερταχείας λειτουργίας του διαδικτύου για την, το θεματολόγιο της ε, ε, ψηφιακής Ευρώπης έχουμε την αρχή ότι έχουμε καλά μελετήσει τα πράγματα, υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν, πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να υλοποιήσουμε αυτή την ανάγκη. Κάθε Ευρωπαίος να έχει δυνατότητα μέχρι το 2013 να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχει μία γραμμή. Είναι σχετικά σύντομα αυτή η ημερομηνία ήδη κοντά μας. Κάθε Ευρωπαίος πρέπει και στις περιοχές της Υπέθρου και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές να έχει δυνατότητα πρόσβησης. Αυτό θα είναι το βασικό πρόγραμμα μέχρι το 2013. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα να κάνουμε για να ανταποκριθούμε ανταποκριθούμε στις ανάγκες των υπηρεσιών. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, ε, συνολική κάλυψη από πλευράς προγραμμάτων και πρέπει να αυξηθεί μέχρι 30 MB ε, ανά δευτερόλεπτο η επίδοση, δίνοντας τη δυνατότητα υπερταχείας σύνδεσης μέχρι 100 MB ανά δευτερόλεπτο το 2020 για πάνω από 50% των πολιτών μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει όχι μόνο με αυτές τις γραμμές αλλά και σε σχέση και με τις ε, γραμμές που θα συνδέονται στην ψηφιακή, στο ψηφιακό θεματολόγιο. Αυτό είναι όχι μόνο το οποίο πρέπει να γίνει, είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι αυτό που πρέπει να επιτευχθεί και μπορείτε με βάση αυτά τα στοιχεία να κρίνετε το τι πρέπει να γίνει. Διαφορετικά, όποιος δεν τα καταφέρει θα είναι υπεύθυνο και θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Έχουμε όμως την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Αν μπορώ να σας δώσω αυτά για να τα μοιράσετε, παρακαλώ. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, ταχύ, ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση. Ευρύ φάσμα επικοινωνία, ευρυζωνικό φάσμα. Και είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι μόνο η ψηφιακή ατζέντα, είναι επίση ε, σε σχέση με την επικοινωνία και αυτή η πτυχή. Θα υιοθετηθεί, θα εγκριθεί υστερότερα εφέτο και ένα κοινό πλαίσιο για να ανταποκριθούμε σε αυτού του στόχου. Θα προτείνουμε φιλόδοξο φάσμα, υπερφιλόδοξο φάσμα που θα ακολουθηθεί και θα παρουσιαστεί μετά τις θερινές διακοπές. Θα επικεντρώνεται στις πολιτικές ε, προτεραιότητες μέχρι το 2015 και θα θέτει σαφέστατους στόχους ε, που θα πρέπει να ε, τηρούνται όσον αφορά την, την υλοποίηση. Ταυτόχρονα θα δώσουμε και μια σύσταση για την πρόσβαση της επόμενης γενεάς για να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές όπως χρειάζεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ώστε να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις στην νέα γενεά ε, ε, ε, στην ψηφιακή Ευρώπη και να ενθαρρυνθεί και ο ανταγωνισμός. Νομίζω μπορείτε να προσυπογράψετε αυτές τις αρχές. Τα συμφέροντα των καταναλωτών και η διασφάλισή τους έχουν κυρίαρχη σημασία. Επίσης, το να αυξήσουμε την δυνατότητα έρευνας στην κοινωνία των πληροφοριών και των τεχνολογιών. Πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις όσον αφορά και τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις για τις επενδύσει να διπλασιάσουμε τις ε, ετήσιες δημόσιες δαπάνες όσον αφορά αυτή την έρευνα σε 11 ευρώ μέχρι το 2020 και θα προτείνουμε και μέτρα για ελαφρότερη και ταχύτερη πρόσβαση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για νέους ερευνητές, καινοτομία μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι αρκετά ενδιαφέροντα για σας ως ιδέες. Θα έλεγα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αρκετά συχνά καινοτόμα θέματα, θέματα καινοτομίας ξεκινούν μέσα στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας μικρομεσαίας επιχείρησης ή επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτούς τους νέους ερευνητές να τους συντάξουμε, να τους συνδέσουμε ώστε να λειτουργούν μέσα σε ένα συντεταγμένο πλαίσιο. Να μην χρειάζονται ατέλειωτα έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται για να μπορέσει κάποιος να τύχει υποστήριξης και θα πρέπει να μπορέσει κανείς να λειτουργεί αμεσότερα και πιο γοργά και πιο αποτελεσματικά. Ολοκληρώνονται δίνοντας το ICT, η κοινωνία της πληροφορίας και των τεχνολογιών και τα ωφέλη που πρέπει να αποβαίνουν προς όφελος των πολιτών. Πολλές ευκαιρίες εδώ χάνονται και πολλά πράγματα πρέπει να δούμε, μεγάλες προκλήσεις, τα θέματα των κλιματικών αλλαγών, οι μεταφορές, πάρα πολλά τέτοια συναφή. Ας υπενθυμίσω κάποιες από τις κυριότερες δράσεις. Να ξεκινήσουμε δουλειά με εμάς τους ίδιους. Έχει νόημα νομίζω να καταδείξουμε ότι εμείς οι ίδιοι συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο που συνάδει Δηλαδή και είναι συμβατός με όλα αυτά ώστε να μπορέσουν άλλοι να ακολουθήσουν το παραδείγμά μας για την χρηστή διακυβέρνηση. Δημόσιες ε, υπηρεσίες που πρέπει ε, στο διαδίκτυο να είναι ε, προσπελάσιμες ε, θα υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα δράσης που θα υιοθετηθεί το 2010 για να αντιμετωπιστούν οι κυριότερες προκλήσεις των επόμενων πέντε ετών. Κινητικότητα στην ενιαία εσωτερική αγορά και περισσότερο φιλικές προς τους χρήστες υπηρεσίες. Ε, μια τέτοια περίπλοκη και σύνθετη ημερήσια διάταξη πρέπει να τύχει σωστής αποτελεσματικής υλοποίησης μέσα από τις σωστές δομές. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη ίδια ευρωπαϊκή Επιτροπής με μια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη πάντα και θα διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ότι οι δικές μας δράσεις θα αντανακλώνται επαρκώς στο επίπεδο των κρατών μελών, στο εθνικό επίπεδο. Και με εσάς θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους σε σχέση με το θεματολόγιο ε, το ψηφιακό θεματολόγιο, ε, διοργανώνοντας ε, ετήσια φόρα όπου θα συνέρχονται τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι εμπλεκόμενοι ώστε να προχωρούν από κοινού. Και θα διασφαλίζουμε ότι θα γίνουν αυτά όπως τα υποσχεθήκαμε στους πολίτες μας και όπως πρέπει. Και φυσικά θα υποβάλουμε έκθεση σχετικά με όλα αυτά στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μόνο δύο-τρία θέματα ακόμα επιπρόσθετα συμπληρωματικά. <clears throat> Θα έχουμε μια έκθεση, ενδιάμεση έκθεση τον Ιούνιο για τις υπηρεσίες περιαγωγής ε, και η σύσταση σε σχέση με τα θέματα περιαγωγής και για ε, την ταχύτητα και το SWIFT ε, και την δυνατότητα να ευθυγραμμιστούμε όσον αφορά την τιμή, τις τιμές υπό τις οποίες το πλαίσιο τιμών καθώς επίσης και ε, ε, τα στοιχεία για την περιαγωγή σε σχέση με το λιανικό εμπόριο και διαφανείς ε, μηχανισμούς. Ένα άλλο θέμα είναι η αμεροληψία και ουδετερότητα. Στο πρόσφατο λόγο που εξεφώνησα κατέστησα σαφές ότι οι, νέοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη δίνουν χρήσιμα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και τα θέματα που αναφύονται. Και επίσης επεσήμανα στον λόγο μου εκείνο ότι θα αποφύγουμε να δώσουμε βιαστικές απαντήσεις. Προτού ε, να έχουμε εξετάσει σε βάθος τα πιθανά ενδυνάμει προβλήματα, αν υπάρχουν κάποια. Δεν είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι, δεν πρέπει με συναισθηματικά φορτισμένο τρόπο να αντιδράσουμε, αλλά αντικειμενικά και νυφάλια. Και έτσι θα ξεκινήσουμε μια σωστή διαβούλευση και εξέταση που θα διοργανωθεί πριν από τις ερηνές διακοπές για να εξετάσουμε να δούμε αν υπάρχει ανάγκη κάποιων πρόσθετων ε, παρεμβάσεων, ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε, επιτρέψτε μου να αναφέρω και πάλι τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσουμε. Ελευθερία της έκφρασης, ε, διαφάνεια, μη διαπραγματεύσιμη και η διαφάνεια. Επενδύσεις σε ένα ανοιχτό δίκτυο πρέπει να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν αθέμητες πρακτικές και να μην υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τους ανταγωνιζόμενους. Και θα υποστηρίξουμε ευκαιρίες στην καινοτομία ώστε να υπάρξουν ε, καινοτόμα πρότυπα. Οι υπηρεσίες μου ήδη ασχολούνται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης ε, για τις ε, οικουμενικές αρχές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων και η διαβούλευση και που βρίσκεται υπό εξέλιξη σε, σχέση, με το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Ένα στοιχείο κλειδί είναι ιδιαίτερα το αν αυτά που προβλέπουμε στην, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος στο τέλος τέλος και μια ανοιχτή ε, διαβούλευση που ολοκληρώνεται και για αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή αναλύουμε αυτές ε, τις ε, διαβουλεύσεις και θέλω να είμαι ειλικρινής και κατηγορηματική τονίζοντας. Ε, δεν έχω κάποια προ, κατηλημένη άποψη ή κάποιες δεδομένες κατευθυντήριες γραμμές το εγχείρημα αυτό δεν μπορεί να εξεταστεί εν κενό. Ξεκινά από, μια, από έναν αριθμό συνδέσεων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών στοιχείων και συντελεστών. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν όλα αυτά να βαίνουν εκ παραλίλου και να αναπτύσσονται σωστά. Είμαι βεβαία ότι οι υπηρεσίες μου, οι εξαιρετικοί υπάλληλοι και συνεργάτες μου εργάζονται άοκνα και θα συνεχίσουν να εργάζονται άοκνα για να μπορέσουν να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις πτυχές ε, μέσα στις διαβουλεύσεις ε, και χαίρονται τη δουλειά που κάνουν και σίγουρα θα καταφέρουν πολλά να πετύχουν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τα κίνητρα και τις πρωτοβουλίες ε, μακροπρόθεσμα για την, την επίτευξη των επενδύσεων και την διασφάλιση ε, εισοδήματος που θα διασφαλιστεί από τους εμπλεκόμενους από αυτές τις επενδύσεις. Και αυτό Επιτρέψτε μου να πω, Πρόεδρε, ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι εκτε να εμπλακούν στο παιχνίδι. Κανένας να μην παραμείνει εκτός ή να μην αγνοηθεί. Θα είναι απαραίτητο να υπάρξει επικοδομητική παρέμβαση, σεβόμενη πάντα ότι ο καθένας έχει τις δικές του ευθύνες, πρέπει όμως να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και στην ανακοίνωση σε σχέση με το ε, φθινόπωρο, Εντοπίζοντα εντοπίζοντας ε, τις ε, διαφορετικές ε, δυνατότητες και εναλλακτικέ λύσεις από πλευράς πολιτικής και τις γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα δράσουμε και επ' και σε αυτό το σημείο ενεργητικά. Έχοντας αναφέρει αυτά, θα ήθελα να ακούσω τώρα τις δικές σας παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ uh, την κυρία Επίτροπο για τη μας παρουσίασε πολλά θέματα και πολύ ενδιαφέροντα γιατί τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με το δικό μας έργο, ειδικά το τελευταίο θέμα. Όπως γνωρίζετε, εγώ ήμουν εισηγητής για την αναθεώρηση του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά έχουμε και το θέμα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την κάρτα με τους στόχους σας. Ε, θα προσπαθούμε να ανταφέρνουμε κοντά μας κάθε φορά που συνεδριάζουμε. Είστε μάλλον η πρώτη επίτροπος ε, που κάνατε κάτι τέτοιο. Ελπίζω να επιτύχουμε τους στόχους μας, ειδικά για την ψηφιακή κοινωνία του 2013. Τώρα, κάθε πολιτική ομάδα θα ήθελα να μιλήσει από μία φορά στην αρχή Προτείνω λοιπόν να έχουμε έναν πρώτο γύρο με... Παρακαλώ κάντε σύντομα σχόλια και ερωτήσεις. Μετά, De Ράπτη, Ζουβάν, Αρίας, Τούν, Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι στις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρώτο γύρο έξι ερωτήσεων και μετά έναν ακόμη γύρο. Αλλά θα πρέπει να κλείσω εκεί τον κατάλογο μιλητών. Θα κάνω και εγώ μια ερώτηση στο τέλος. Ο κύριος Σουβάμπ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για αυτή την κάρτα. Είναι ένα παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης ε, σκέφτηκα ότι κάποιο iPad θα μας δίνατε, ε, αλλά πρέπει να εξοικονομήσουμε βέβαια και αυτό είναι το δώρο που μας κάνετε εσείς. Λοιπόν, εντάξει, η πρώτη μου ερώτηση καταρχήν. Καταρχήν θέλω για αυτό το περιεκτικό έγγραφο και που εγκάρσια μεταξύ των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμφωνηθεί να σας ευχαριστήσω. Είναι πραγματικά πολύ φιλόδοξο. Και όταν σας λέω ότι στους στόχους που θέλετε να επιτύχετε σε αυτούς θα μετρηθείτε, με αυτούς θα μετρηθείτε, αυτό είναι θετικό. Μακάρι να καταφέρετε να επιτελέσετε πολλούς από αυτούς, το δυνατόν περισσότερους. Εγώ ίδιο θέλω να θέσω κέντρο βάρους σε τέσσερα τέτοια θέματα όπου προτείνεται μέχρι το 2012 να υπάρξει ένα, η επιλογή ενός ε, ε, ε, εθελούσιου πλαισίου για αυτή την πρόθεση. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή με μεγάλη προσπάθεια εργοδός θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε αλλά να μην είμαστε αφελείς. Δεν θα είναι απλό το εγχείρημα. Και αν τα βλέπουμε σωστά τα πράγματα υπάρχει πολιτική βούληση εδώ που αντανακλάται σε αυτό το έγγραφο. Ίσως όμως πρέπει να μην ξεχνάμε τα κράτη-μέλη που και αυτά θα πρέπει να άλλη πλευρά να διαβουλευτούν και να προχωρήσουν. Δεύτερον, η σύγκριση της Ευρώπης με της ΗΠΑ στον τομέα online. Είναι σαφής η σύγκριση στα αποτελέσματά της. Έχουμε και διαφορετικέ αλλαγές όμως, διαφορετικούς όρους. Στις ΗΠΑ στον τομέα online έχουμε τελείως άλλες δυνατότητες ανάκλησης Όλα αυτά με ένα δικαίωμα μιας κάρτας λειτουργούν και δεν είναι ανάγκη ο, ο πάροχος ή ο έμπορος να ε, είναι ο διαμεσολαβητής αλλά ε, ο πάροχος της ε, κάρτας, της πιστοτικής κάρτας με την οποία αγοράζει ο καταναλωτής. Πρέπει λοιπόν κάπως πιο ρεαλιστικά να υπολογίζουμε και αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Δεύτερο σημείο, περαιτέρω εξέλιξη μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο εμπόδιο να αγοράζουν οι πολίτες στην Ευρώπη online ηλεκτρονικά είναι η γλώσσα. Αλλά το δεύτερο σημαντικότερο εμπόδιο στα νομικά θέματα είναι η ε, διεξαγωγή, η διασφάλιση των πληρωμών. Θα έπρεπε να κάνετε προσπάθεια να μπορούν αυτές οι πληρωμές να γίνονται μέσα σε τακτά πλαίσια και μέσα σε γοργότερες προθεσμίες. Ευχαριστώ. Uh, thank you very uh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέπαρ, Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και εσάς πολύ κυρία Επίτροπε για την πραγματικά πάρα πολύ καλή ε, παρουσίαση και αφομοίωση παρουσίαση αυτών των στοιχείων. Και εγώ το είχα σκεφτεί ότι κάτι συγκεκριμένο χειροπιαστό πια υποβάλλεται επί τραπέζης με το οποίο μπορεί να δουλέψει κανείς ως βάση. Και το χαιρετίζω πολύ αυτό. Και υπάρχουν τόσες πολλές δράσεις που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά επέλεξα μόνο τρεις από αυτές τις δράσεις. θα ήθελα να εμβαθύνω σε αυτές. Το ένα είναι και η πρωτοβουλία υπαριθμών 4, όπως ανέφερε και ο κύριος Σβάμπ. Είναι συγκυρία το ότι ε, συμπίπτει αυτή η επιλογή μεταξύ μας. Είπατε ότι θα πρέπει να εξετάσετε τα νομικά πλαίσια και την δυνατότητα υποστήριξης. Είναι σημαντικό αυτό για την εμπιστοσύνη των πολιτών να την καλλιεργήσουμε διασυνοριακά, να δούμε πώς ένας πολίτης θα μπορεί να διασφαλίζει τα δικαιώματά του. Και είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το χαιρετίζω το ότι κατευθύνεστε προς αυτή την κατεύθυνση και θέλετε εκεί να οδεύσετε. Και πολύ γοργά πρέπει να προχωρήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το δεύτερο κέντρο βάρους για την δράση που θα ήθελα να επιλέξω είναι η παριθμόν 10. Έχω μία ερώτηση σε σχέση με αυτήν. Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω και πάρα πολύ δύσκολη στην επίτευξη και ολοκλήρωση δράση, δράση κλειδί. Θα ήθελα να ρωτήσω μια και πρόκειται και για τις αρμοδιότητες των παραδοσιακών χρηστών που πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο τους και να ε, δράσουμε σωστά. Ξέρετε ότι για την αναγνώριση επαγγελματικών ε, ε, πτυχίων είναι σημαντικό μια προσέγγιση στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να είμαστε ταχύτεροι από τις κράτη-μέλη και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα ή τα προσκόμματα όταν εθνικά διπλώματα ή πτυχία έχουμε μπροστά μας που πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία και θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου να καταφέρουμε να προχωρήσουμε πολύ μπροστά με ένα ας το πούμε κοινό πρότυπο ή διαβατήριο. Επίσης για την δράση κλειδί υπαριθμών 12 κοινέ μέθοδοι για την μέτρηση της ε, ενεργειακής ε, αποδοτικότητας. Είναι πραγματικά κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ λίγο το συζητάμε αυτό. Όταν κάνουμε λόγο για μηχανές, ε, για παράδειγμα ψαχτήρια, ψαχτήρια στο διαδίκτυο, δεν είναι πολύ ακριβό για τον επιμέρους χρήστη αυτό. Όμως, όταν είναι μεγαλύτερων διαστάσεων. Έχουμε μεγάλες μηχανές, μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούν, καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ε, ένταση ενέργειας, ε, πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το θέμα για να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Ε, Κύριος Κρότσμαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω Έχετε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, κυρία Επίτροπε. Είδα την κάρτα σας. Είναι εξαίρετο αυτό που μέχρι το 2015 θέλετε να πετύχετε και δεν είναι και τόσο μακριά το 2015. Πολλά θέλετε να κάνετε λοιπόν. Όταν ξέρουμε ότι 30% το αναφέρατε στις εκθέσεις σας, σήμερα δεν χρησιμοποιούν καν το διαδίκτυο. Και μέχρι το 2015 50% να θέλετε να καλύψετε από πλευρά των πολιτών μας είναι εξαιρετικό πράγμα. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν την πρότασή σας και τις προσπάθειές σας. Είπατε στην έκθεσή σας ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη από πλευράς καταναλωτών. Εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο και στην ασφάλεια και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Χρειαζόμαστε και προσπελασιμότητα και ταχύτητα και αύξηση του βαθμού βαθμού εκμετάλλευσης. Όλα αυτά που θέλετε να πετύχετε είναι και θέματα της Επιτροπής μας για, που έχουμε εξοικειωθεί με θέματα προστασίας των καταναλωτών. Έχουμε το ψηφιακό θεματολόγιο. Σίγουρα θέλουμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε όλους τους στόχους σας. Έμαθα ότι οι στόχοι μπορούμε, μπορούν να πετυχαίνονται μόνο όταν οι άλλοι από τους οποίους εξαρτώμαστε συνεργάζονται για την επίτευξή τους και αυτοί. Έχω υπόψη μου σε σχέση με την περιαγωγή του 2009 που έδωσε προτερήματα για τους πολίτες έγινε χειροπιαστή και μπόρεσε να αναγνωρί... μπόρεσαν οι πολίτες να αναγνωρίσουν ένα συμπαθητικό θελκτικό πρόσωπο της Ευρώπης. Τώρα σε σχέση με την κατάσταση των, ε, ε, της περιαγωγής σήμερα πού θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη δράσης για την περιαγωγή, το roaming στο μέλλον. Θα μπορούσε ένας κανονισμός roaming 3, περιαγωγής 3 να επιτευχθεί για να σημειωθούν περαιτέρω γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ χειροπιαστό και ε, ξεχωριστό και εδώ τα προτερήματα της Ευρώπης ως πλεονεκτήματα θα είναι σαφή για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Άγκστρομ παρακαλώ στην συνέχεια. Thank you. Ε, well, the... Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για την ενημέρωση πολύ θετική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή στο μέλλον. Τώρα, αρκετά θέματα που θέλουμε τουλάχιστον σταδιακή αναθεώρηση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να υπάρξει εξυγχρονισμός. Άλλο θέμα, η ιδιαιτερότητα του δικτύου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ίσως χρειαστεί κανονισμός κατά τη γνώμη μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το συζητήσουμε. Περιαγωγή δεδομένων, το ανέφερε και ο κύριος Κρόιτσμαν. Αυτή τη στιγμή δεν επουφελόμαστε των νέων τεχνολογιών όταν πρέπει να πληρώσουμε χιλιάδες ευρώ για να χρησιμοποιήσουμε περιαγωγή δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε άκουσα πολλά θετικά και χαίρομαι γι' αυτό. Μία ερώτηση για την δράση 5 διαλειτουργικότητα και πρότυπα. Πρόκειται για θέματα πολύ σημαντικά. Όμως υπάρχουν πολλές ανησυχίες εντός των χρηστών του διαδικτύου γιατί Υπάρχει μία φήμη ότι αρχικά ο τίτλος ήταν «Διαλειτουργικότητα και ανοιχτά πρότυπα» και μετά διαγράψατε το «ανοιχτά». Όπως είπατε, πολλή καινοτοπία έρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η διαφορά μεταξύ καθαρά ανοιχτών προτύπων και σχετικά ανοιχτών προτύπων σχετικά χρήσιμων προτύπων είναι πολύ μεγάλη. Γιατί κάποιες χιλιάδες ευρώ μπορεί να μην είναι τίποτα για μια μεγάλη εταιρεία, αλλά για μια μικρομεσαία επιχείρηση είναι η διαφορά που θα τους ε, κάνει να ασχοληθούν με το θέμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά τα ανοιχτά πρότυπα και μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, γενικά αναμένουμε με ανυπομονησία τις πρωτοβουλίες σας. Κυρία Μακλάρκεν, Ευχαριστώ την ε, Επιτροπό για τα σχόλια της ε, και για την αποφασιστικότητά της. Για την ε, δική μου περιφέρεια τα East Midlands που ακόμη περιμένουν να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση είναι πολύ σημαντική η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να υπάρξει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ρωτώ λοιπόν πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια όσο το δυνατόν ίση πρόσβαση στο ίντερνετ. Και επίσης για το 2013 δεσμεύεστε για μια βασική ευρυζωνική σύνδεση. Πώς θα το κάνετε αυτό. Και χρειάζεστε και κάποια συνεργασία με τους μεγάλους παίκτες οι οποίοι πρέπει να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις ευρυσονικές συνδέσεις. Από την άλλη πλευρά όμως πιέζουμε αυτή τη στιγμή τους προϋπολογισμούς. Πώς θα τα καταφέρουμε. Κύριε Τρεονταφυλλίδη παρακαλώ. To thank the Commissioner for uh, presenting her program such uh, clarity. Να ευχαριστήσω την Επίτροπο που με τόση σαφήνεια παρουσίασε το πρόγραμμά της. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και αναρωτιέται κανείς αν θα τα καταφέρουμε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Της εύχομαι κάθε επιτυχία. Αναμένω με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των δημόσιων διαβουλεύσεων, ενδεχομένως και με συμμετοχή του Κοινοβουλίου, γιατί πρόκειται για θέματα που αφορούν τις ζωές όλων των πολιτών. Αναμένουμε λοιπόν όλες τις πρωτοβουλίες σας και θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στο έργο σας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Μας μένουν 20 λεπτά. Θα απαντήσει τώρα η Επίτροπος και να προτείνω κάτι για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ένα λεπτό ο καθένας σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε για τα ερωτήματα και ξεκινάω εγώ πρώτος για να σας δώσω το καλό παράδειγμα. Έτσι θα κάνουμε σε 10 λεπτά τις ερωτήσεις και θα έχει 10 λεπτά για απαντήσεις η Επίτροπος. Ξεκινάω λοιπόν εγώ. Ένα λεπτό. Ήθελα να σας ρωτήσω κυρία Επίτροπε το εξής. Τονίζετε το ότι θα μας ενημερώσετε για τον κανονισμό για την περιαγωγή. Όμως στην οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες και τα δικαιώματα του καταναλωτή υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και για την περιαγωγή. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα εξής. Καταρχάς, δυνατότητα μεταφοράς του αριθμού κινητού τηλεφώνου άμεσα. Δεύτερον, οι περιορισμοί στους όρους των συμβολέων. Τρίτον, προσυμβατική ενημέρωση και προδιαγραφές ποιότητας. Τέταρτον, προδιαγραφές για τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα ασχοληθείτε τόσο πολύ με τα δικαιώματα αυτά των χρηστών όσο και με την περιαγωγή. Γιατί έχουμε τονίσει πολύ το απεριαγωγή, ενώ υπάρχουν και άλλα θέματα εξίσου σημαντικά. Κορεχάντε Κάμπος. Uh, uh, Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στις δημόσιες συμβάσεις ως ε, θέμα όπου θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά κενά και χρειάζεται νομοθεσία. Όντως, οι δημόσιες προμήθειες είναι πολύ σημαντικές και θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο οι ηλεκτρονικές ε, προμήθειες. Υπάρχει και άλλο θέμα, οι καθυστερημένες πληρωμές του δημοσίου. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια, τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, ε, την ε, μείωση των στρεβλώσεων της αγοράς και τη μείωση του κόστους ε, και για τους ε, αγοραστές ε, και για τους προμηθευόμενους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν πρόκειται να ξεκινήσετε μία πλατφόρμα φέτος ή κάποια νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές υποβολές προσφορών. Κύριε Ράπτη. Επίτροπε για την εισήγησή σας. Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω πότε νομίζετε, πότε προβλέπετε ότι θα μπορούμε να έχουμε έναν αριθμό τηλεφώνου στην Ευρώπη για όλα τα κράτη. Δεύτερον, αν θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τις οριζόντιες συνεργασίες που έχετε με συναδέλφους σας, δεδομένου ότι όλα αυτά που μας είπατε αγγίζουν πάρα πολλούς τομείς και άρα πάρα πολλές πολιτικές. Και τρίτον, να σας ευχαριστήσω για αυτή εδώ την κάρτα, ε, γιατί δείχνει πέρα από όλα τα άλλα ότι είστε και πάρα πολύ θαραλέα. Γιατί διότι αυτή την κάρτα χαρήκαμε όλοι που την πήραμε σήμερα, αλλά θα την έχουμε κοντά μας ως το 2014. Και εκεί που θα ξανάρθετε ε, θα κοιτάμε τους αριθμούς και θα ρωτάμε να μας πείτε τι έχετε επιτύχει. Ευχαριστώ. Perfect timing, Mrs. Thank you. And Ακριβώς το χρόνο, κυρία Ράπτη. Και να πω ότι και εγώ έχω βάλει στη λίστα μου αυτό που αναφέρατε για τον μοναδικό αριθμό τηλεφώνου. Κύριε Μάντερς, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για το φιλόδοξο σχέδιό της πάντα είναι υψοκίνδυνο το να μας δίνετε προθεσμίες και να τις γράφετε και σε μία κάρτα γιατί θα μπορούμε να τα ελέγξουμε μετά. Ελπίζω όμως ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες σας. Αυτό πάντως που δεν είδα, γιατί μιλάμε εδώ για εργαλεία στο τομέα ICT, αλλά αυτό που δεν είδα, που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αν και δεν συνδέεται άμεσα με τη δική μας Επιτροπή, μόνο έμεσα, είναι η ηλεκτρονική μάθηση, που είναι το μέλλον. Δεν τα καταφέραμε με τους στόχους της Λισαβόνας για να γίνουμε η πιο ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης παγκοσμίω, αλλά ελπίζω ότι θα κάνετε κάτι κατά τη διάρκεια της θητείας σας για το θέμα της ηλεκτρονικής μάθησης. Μετά, σημείο δράσης 9, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Γνωρίζω ότι θα ασχοληθείτε με το θέμα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μειώσετε και την γραφειοκρατία εδώ. Γιατί συνήθως όταν έχουμε μια καλή πρωτοβουλία, αλλά εξαιτίας της γραφειοκρατίας δεν καταφέρουμε να επιτύχουμε τους πραγματικούς μας στόχους. Ελπίζω ότι η ψηφιακή σας ατζέντα θα μπορέσει να κάνει κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριο Ζουβάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί κειμένου της ε, Επιτρόπου είδαμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους, οπότε και εγώ θα κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Χρησιμοποιείτε τον όρο διανοητική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία. Και μιλάτε και για συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρώπη είναι ένας γεωγραφικός χώρος που βασίζεται στον πολιτισμό και στην διανοητική προστιθέμενη αξία. Αν λοιπόν δεν προστατεύσουμε την διανοητική ιδιοκτησία, τότε αλλάζουμε κάτι στον πολιτισμό μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν θέμα η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεύτερον, λέτε καλώς ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο χρόνο για να ακούσουμε πριν κάνουμε προτάσεις. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για την ουδετερότητα του δικτύου. Είπατε ότι είναι σημαντικό θέμα, συμφωνώ, αλλά δεν μου αρκεί αυτό για να καταλάβω προς τα που θέλετε να κινηθείτε. Ο κύριος Αρίας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ σήμερα για να μας πείτε ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας σε σχέση με την ψηφιακή θεματολογία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι για τα 200 300 ερωτήματα δεν υπάρχει χρόνος για να τα διατυπώσω, μια και αυτά είχα υπόψη μου. Αλλά να πω απλά ότι στεναρά πιστεύω ότι έχετε στα, χαρτιά σας το πιο, στα χέρια σας το πιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να θα προχωρήσετε την ψηφιακή Ευρώπη. Πρέπει να προλιάνουμε το έδαφος για τις μελλοντικέ γενναίες, όχι για μας αλλά για τους ε, επόμενους. Κάποιοι από εμά έζησαν αυτήν την επανάσταση, οι άλλες γενναίες θα ζήσουν 100% όμως μέσα στο πλαίσιο αυτής της νέας ψηφιακής εποχής και αυτής της επανάστασης στα ψηφιακά που ζούμε πρέπει να σκεφτούμε και να συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε για αυτή την ε, επανάσταση την ψηφιακή του τι σημαίνει και το τι θα συνεπάγεται και το βλέπουμε ήδη σήμερα και να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για να μπορέσει να ανταγωνιστεί μέσα στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής. Τούτου λεχθέντος δεν μπορώ να επικεντρωθώ σε 200 ή 300 ερωτήματα, σε ένα. Είναι πολύ απλό. Για τα δίκτυα στο μέλλον που θα ζήσει αυτή η νέα γενεά πιστεύω ότι πολύ σημαντικό θα ήταν να δημιουργήσουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι ε, σημαντικό ε, στοιχείο. Είναι μια γενεά που είναι καταδικασμένη εντό εισαγωγικών να ζήσει αυτή την ψηφιακή εποχή. Ένα από τα θέματα τα πιο σημαντικά είναι η παιδεία, η εκπαίδευση. Να εκπαιδεύσουμε, να παιδεύσουμε αυτή τη νέα γενεά ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί και να εξοικειωθεί στα ψηφιακά. Θα ήθελα να ακούσω τι απόψει σα σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τέλος κυρία Τούνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι Κάθε φορά που βλέπω τον τηλεφωνικό μου λογαριασμό θεωρώ ότι όσοι ταξιδεύουν είναι αποκομμένοι από την ηλεκτρονική ενημέρωση. Κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Μας μιλήσατε για φορητότητα του τηλεφωνικού αριθμού και για τις μηδενικές χρεώσεις για την περιαγωγή. Πρόσφατα συζητούσα το θέμα με υπαλλήλου της ε, France Telecom και μου έλεγαν κάτι για, μία, για έναν ευρωπαϊκό αριθμό τηλεφώνου. Νομίζω ότι θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Τι ακριβώς πιέσεις πρόκειται να κάνετε στα κράτη-μέλη για να επιτύχετε τους στόχους σας. Για να μην είναι το τηλέφωνο από Βέλγιο σαν να είναι προς τη Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστούμε. Έχετε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή σας κύριε Επίτροπε. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε σε το δυνατόν περισσότερα πράγματα αμέσως. Ευχαριστώ. Um, uh, Αρκετά μεγάλη πρόκληση και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εκδήλωση της Ισπανικής Προεδρίας. Διοργάνωσε η Ισπανική Προεδρία μια πλατφόρμα με 800 νέους ερευνητές. Είχαν προσκληθεί να πάνε στη Μαδρίτη αυτοί οι νέοι και αρνήθηκαν να πάνε σε ξενοδοχεία. Πήγανε σε αντι... Είχαν κάποιε σκηνέ αντίσκηνα όπω τα αποκαλούσαν. Πήγαν εκεί με του υπολογιστέ του, βγαίνανε με του υπολογιστέ του, συζητούσαν, είχαν επαφέ και διαλόγου με όλου του ε, ενδιαφερόμενου ε, και έτσι ήταν. α το πω έτσι, υπήρχαν τμήματα παραγωγική ε, ψηφιακή δράση. οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και εμεί περπατούσαμε εκεί και κάποια στιγμή κάποιος βρισκόταν εκεί πιο ψηλά από τους άλλους και οι άλλοι ε, από τους 800 ας το πω έτσι καθόντουσαν γύρω και διατύπωναν ερωτήσεις και ρώτησα μα ποιος είναι αυτός εδώ δεν τον αναγνωρίζω ποιος είναι ο κύριος και κάποιοι από την αντιπροσωπεία μου μου είπαν είναι ο κύριος Χίψη και είπα δεν έχω ιδέα ποιος είναι εκείνος είδε ότι εγώ ρωτούσα όμως και είπε είμαι ο Χί ο έκανε τις, ε, αυτό συστήθηκε ήταν όμως μεγάλος ήρωας για αυτούς τους νέους που είχαν συναθριστεί εκεί. Και είπε, μα εσείς είστε ακόμα από τη γενιά του Bill Gates και του Steve Jobs, έτσι, είπε στους δικούς του, κοιτάξτε πίσω σας, εκεί υπάρχει μια αντιπροσωπεία, είναι η προηγούμενη, η παλιά γενναία. Και αν και δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι πρέπει να γίνει και τι ε, πρέπει να γίνει. Αν δεν ξέρουν τι πρέπει να γίνει θα είμαστε εμείς η χαμένη γενιά, η χαμένη του μέλλοντος. Και στη συνέχεια συζητούσαμε, όχι με όλους αυτούς τους 800, αλλά με κάποιους. Ο νεότερος ήταν 14 ετών παρακαλώ. Ένας νέος 14 ετών. Είχε τρεις πατέντες ήδη καινοτομία. Είχε ξεκινήσει δύο επιχειρήσεις αυτός ο 14 χρονος Και συζητώντα με όλα επί παντός του επιστητού. Αυτό το οποίο ήταν το πιο θελκτικό και εντυπωσιακό ήταν ότι συζητούσαν με, τις, με τους υπολογιστές τους και έδειχναν ένα στον άλλο την οθόνη και τον υπολογιστή του και Είπα, μα τρελό είσαστε, εξηγείτε την πατέντα σα και την επινόησή σα στους άλλου. Και είπε, γέλασε, μα δεν καταλαβαίνετε. Α, συνεργαζόμαστε, αυτό είναι το πιο θελκτικό για μα. Δείχνει ο ένα τον άλλο την έρευνά του. Εμεί έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο και γι' αυτό ακριβώ ο κόσμο και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο με την συνεισφορά όλων των άλλων που συμμετέχουν. Αυτό είναι περί του οποίου πρόκειται. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η νέα γενεά δρά, με αυτόν τον τρόπο είναι διαφορετική από τους άλλους αυτή, είναι η γενεά που πρέπει να μας κάνει να δούμε και να καταλάβουμε τι πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αυτό έγινε. Και μία από τις ιδέες που είχα και σε αυτήν εργαζόμαστε είναι να μπορέσουμε σε σχέση με καθηγητές και επαΐοντες ως συμβούλους, να καταλήξουμε με ένα ευρύτερο τέτοιο πλαίσιο συμβούλων, ώστε να ενταχθούν οι δυνατότητες και οι καινοτομίες για αυτούς τους νέους μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα σας ενημερώσω για αυτό το στόχο αυτής της μονάδας. Αλλά δεν είμαστε πια εμείς ή κάποιοι που θα μάθουν εκείνους κάτι, εκείνοι θα μας μάθουν εμάς και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε. Τούτου λεχθέντος Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε. Είμαστε φιλόδοξοι, υπάρχει φιλοδοξία, υπάρχουν ζητήματα και ξέρουμε ότι αυτά δεν είναι τίποτα το καινούριο, όμως τούτων λεχθέντων εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα να κάνουμε λόγο για ε, ασφάλεια, για την παιδεία, εκπαίδευση. Ο γενικότερος στόχος γι' αυτό είναι να δούμε αυτό το πλαίσιο. Τι πρέπει να κάνουμε. Είμαι πρόθυμη να ακούσω οποιαδήποτε δική σας συνεισφορά και πρόταση. Ο χώρος ενιαίων πληρωμών και ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών. Ήδη είχαμε εμπλακεί και εργαζόμαστε ως προηγούμενη ε, επιτροπή για αυτό το θέμα. Συμφωνώ, είναι μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε συγκεκριμένα σε αυτή την πορεία, καθορίζοντας μια ημερομηνία για τη τις διαπραγματεύσεις, για τις διαβουλεύσεις. Μετά, προστασία προστροπικών δεδομένων, προστασία δεδομένων. Η συνάδελφος κυρία Ρέντινγκ προγραμματίζει, σχεδιάζει μια αναθεώρηση και πρέπει από κοινού εκ παραλίλου να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε και να συντονιστούμε πρέπει να έχουμε σαφείς βελτιώσεις. Και αυτό πήρα ως μήνυμα από εσά. Παρακαλώ να ε, διασφαλιστεί η βελτίωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τις δράσεις κάνω λόγο τώρα. Είμαι πρόθυμη να υποβάλω προτάσεις επινομικών μέτρων και μέσων αν στον τομέα του ICT, της ε, κοινωνίας των πληροφοριών και των τεχνολογιών, ε, αν υπάρχει ανάγκη να αναλυθεί δράση. Για παράδειγμα, όσον αφορά και τα ε, θέματα της, των, της επίδοσης στα ενεργειακά. Πρέπει να είμαστε σε θέση και ικανοί να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτή την ε, ψηφιακή θεματολογία. Αυτό είναι αυτό το οποίο είναι το διακύβευμα, το στίχημα. Αυτό είναι το μεγάλο άλμα. Να πάρουμε το θέμα της περιαγωγής δεδομένων. Αν δεν είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να συμπεριλάβουμε όλα τα οποία συνδέονται, διότι όλα συνδέονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε αυτά τα θέματα περιαγωγής δεδομένων και σε σχέση με τη δική μου εμπειρία και βιώματα και από την προηγούμενη πείρα, αν πρέπει κανείς να, διαπραγματεύει, να διαπραγματεύεται κάτι, αν επιλέγει το ένα ή το άλλο και λέει τούτο πρέπει να επιληθεί τώρα, αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Αυτό δεν είναι η εξέβρεση λύσεων για το σύνολο, για ένα ευρύτερο σύνολο. Εμείς συνειδητοποιώντας αυτό που πρέπει να γίνει, και αυτή είναι η γραμμή που ακολουθώ, πρέπει να εντάξουμε όλα τα κομβικά στοιχεία, όλα τα, όλους τους συντελεστές σε ένα πλαίσιο επιτραπέζης και να συνέλθουμε γύρω από αυτό το τραπέζι με όλους τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους. Ε, και δώστε μου μια ευκαιρία παρακαλώ, ακούω τις παρεμβάσεις σας, ε, συνειδητοποιώ πώς εσείς ε, ευαισθητοποιείστε και αντιδράτε σε σχέση και με τους ε, ψηφοφόρους σας και τα θέματα που τους αφορούν. Είναι ένα από αυτά τα θέματα λοιπόν αυτά, όπου είμαι πρόθυμη και έχω η ίδια αυτή την πείρα, ακούω τις απόψεις και σε σχέση με την, τον έναν ή άλλο τομέα με ρωτάνε πράγματι είναι η ψηφιακή αγορά αυτή, αν είναι η ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά, αυτά τα οποία μας εξηγείτε, τότε πώς μπορείτε να επεξηγήσετε ότι μπορώ να αγοράσω ένα CD σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, αλλά downloading, να ε, κατεβάσω από τον υπολογιστή μου κάτι, δεν γίνεται αυτό ανεμπόδιστα, απρόσκοπτα παντού. Πρέπει να υπάρξει και κάποια πληρωμή. Και... Λοιπόν, είναι σαφές εδώ ότι οι πολίτες δεν είναι ακόμα πρόθυμοι να πούν εντάξει αγοράζω πολλό, όλα αυτά στο διαδίκτυο γίνονται, θα γίνονται όλο και περισσότερο και θα ευνοούνται περισσότερο. Πρέπει να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια αγορά, αλλά είναι και παράνομη. Ε, ως πολιτικοί όταν γνωρίζουμε ότι κάτι είναι παράνομο πρέπει να αναλάβουμε αμέσω δράση να το αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς χάνουμε την αξιοπιστία μας και καταβαραθρονόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα πράγματα αν δεχόμαστε την παρανομία και δεχόμαστε μια τέτοια έκρηθμη κατάσταση. Κάνοντας λόγο λοιπόν για την ρύθμιση των θεμάτων περιαγωγής και την προσωρινή ε, διάμεση έκθεση θα επανέλθουμε σε εσά και ήδη εφέτος ε, θα έχουμε την πρώτη αναθεώρηση κατά το θέρος και θα δώσουμε μηνύματα για το τι πρέπει να γίνει. Μην θεωρήσετε ή συμπεράνετε ότι όταν καταλήγουμε σε κάποιο αποτέλεσμα αυτό το καλοκαίρι θα σταυρώσουμε, θα σταυρώσουμε τα χέρια μας και θα πούμε «Ε, δεν θα κάνουμε τίποτα με το 2011, δεν είμαστε αφελείς, δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε προσπάθειες και θα αναλαμβάνουμε δράση όπου θα είναι αναγκαίο και όταν κάτι διακυβεύεται για να είμαστε αποτελεσματικοί. Οι ανοιχτές προδιαγραφές τώρα. Είναι σωστό το ζήτημα αυτό. Και ποτέ σε σχέση με ε, ε, διαρροές ε, ή άλλα αντίστοιχα θέματα δεν υπήρξε κάποιο μείζον θέμα. Δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι είναι τέλεια όλα. Είναι αληθεύει ότι υπάρχουν προβλήματα. Όμως αν είναι μόνο η ένας αγώνας για ένα επιμέρους θέμα, θα μπορούσε κανείς να πει Κοιτάξτε, έχουμε περισσότερα θέματα και πιο σημαντικά να ασχοληθούμε. Γι' αυτό δέχομαι και γι' αυτό έρχομαι με αυτές τις ε, προτάσεις και με αυτόν τον τρόπο. Να είναι σαφές ε, ότι έχω και κάποια ιστεροφημία και πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Διαλειτουργικότητα και ανοιχτές ε, προδιαγραφές. Από το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο που είχα για τον ανταγωνισμό είναι σαφές ότι πρέπει να πω ότι αυτά είναι σημαντικά θέματα. Το περιεχόμενο λοιπόν εδώ αυτού του χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να είναι ε, σημαντικό για μένα και είμαι προβλέψιμη στις ε, απόψεις και τοποθετήσεις μου. Δεν πρόκειται να βρεθεί κάτι απροσδόκητο, απρόσμενο μπροστά σας. Χρειαζόμαστε αυτή τη δράση. Χρειαζόμαστε ευρύτερη πρόσβαση για όλους. Με μια ανοιχτή στρατηγική ε, να είναι δυνατή η δράση μας, μπορούμε να βρούμε τη σωστή ορολογία και να καλύπτεται και η σωστή δράση και συντονισμός με τα κράτη-μέλη. Και την εξέβρεση επενδύσεων όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είχαμε επαφές και συζητήσεις με την ΕΤΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ενδιαφέρονται και εκείνοι. Η σύσταση NGA, το ε, ευρυζωνικό φάσμα και το εγχείρημα για το φάσμα συνολικά ε, Spectrum στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φτάσουμε σε κάθε πολίτη. Για να φτάσουμε σε κάθε πολίτη έχουμε ξεκινήσει μια έκθεση στα κράτη-μέλη με αντίστοιχη παρουσίαση μέσω πρέσβεων. Πρέπει να περάσουμε διασυνοριακά και να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται στους πολίτες μας. Και όταν λέω και θέλω να το επαναλάβω αυτό, κάθε Ευρωπαίος πρέπει να έχει δυνατότητα ε, πρόσβασης ε, στο διαδίκτυο και να έχει μια τέτοια σύνδεση είτε ζει στην επαρχία είτε σε απομονωμένη περιοχή ε, στην Ήπεθρο είτε σε νησιά να μπορεί να έχει τη δική του σύνδεση και θα πρέπει να μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε ώστε να είναι οι όροι του παιχνιδιού θεμητοί και δορυφορικά να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά και να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες. Εκεί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εν παρόδο και την αναθεώρηση των οδηγιών, για, της οδηγίας για τις επιχορηγήσεις, κρατικές ε, ενισχύσεις ε, για να μπορέσουμε να αποτροχοπεδίσουμε τα πράγματα. Ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Χάμπορ, είχε διατυπώσει ένα ερώτημα που στενά συνδέεται με την ψηφιακή θεματολογία. Εμείς εκείνο που εμπνεόμαστε 100% να δράσουμε είναι υπέρ των πολιτών. Οι πολίτες ποιοι είναι, είναι καταναλωτές. Είναι 500 εκατομμύρια καταναλωτές για τους οποίους αγωνιζόμαστε. Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι λοιπόν οπωσδήποτε ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των καταναλωτών στο ψηφιακό θεματολόγιο, κάνοντας λόγο και για θέματα υγείας με τον συνάδελφο Ντάλι. Θα βοηθήσουμε να επικεντρωθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Είμαστε γνώμονες σε εσά. Είσαστε ξεκάθαροι στις ε, τοποθετήσεις. Δεν υπήρχε τίποτα το ε, ακατανόητο. Σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν παρανοήσεις ότι θα προχωρήσουμε με τρόπο ώστε να υπάρχει καλή συνεννόηση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και ένα πολιτισμικό στοιχείο στις, ε, <laughs> στην επαφή μας αυτή. Τώρα, ευρωπαϊκό ε, δίκτυο ε, στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσω την πρότασή σας. Ακούγεται θελκτική. Προτού πω ας το κάνουμε και ας ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση και μετά με κατηγορήσουν κάποιοι ότι δεν το είχα σκεφτεί και ότι βιαστικά αποφάσισα κάτι, θα το ξαναδούμε. Θα το συζητήσω με τους συναδέλφους μου επιτρόπους και θα επανέλθω να σας πω τα σχετικά. Αφ' αυτού θα ήταν κάτι ωραίο αν μπορούσε να γίνει. Κάτι καλό που θα μπορούσε να προαχθεί δεν θα, λέγα, θα ανέφερα τώρα ε, ονομαστικά. Αναφέρατε την ηλεκτρονική εκπαίδευση και μάθηση. Η κατάτηση και εκπαίδευση είναι σημαντικό στοιχείο. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει και με θέλγει δεν είναι ότι 30% του πληθυσμού είναι παρθένο σήμερα, δηλαδή δεν έχει εξοικειωθεί και δεν έχει ελογιμότητα ψηφιακή, δεν έχει μάθει τα στοιχειώδη σε σχέση με την ψηφιακή ε, τεχνολογία. Αλλά το 38% θα έπρεπε να μειωθεί σε 15% και πάλι θα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό που δεν θα έχουν εξοικειωθεί με αυτή την τεχνολογία. Αυτό που θέλω να πω είναι αν υπάρχει απουσία εκπαίδευσης ή παιδείας σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να δούμε όχι μόνο ότι υπάρχει αυτό το 30% που θα πρέπει να μειωθεί σε 15% κτλ. Πρέπει να δούμε εκείνους που ήδη σήμερα εμπλέκονται στις ψηφιακές δράσεις, αλλά είναι μια διαδικασία διαβίου μάθησης και εκμάθησης. Οι νέες εξελίξεις και τα νέα στοιχεία ακόμα και στους δικούς μου ανθρώπους ε, που όταν ε, ε, έχουμε κάποια επαφή σε σχέση με θέματα τεχνολογίας, ε, έρευνας, ανάπτυξης, τα πράγματα πάνε τόσο γρήγορα που δεν μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει ανεμπόδιστα. Πρέπει διαβίου να μαθαίνει κανείς και να εξοικειώνεται. Αλλιώς χάνει τις ευκαιρίες. Εκπαίδευση, παιδεία. Αν δεν υπάρχει εκπαίδευση, παιδεία, δεν μπορεί να αναμένει κανείς οι πολίτες να βρουν το δρόμο του σωστά και να υπάρχει και εμπιστοσύνη στην ψηφιακή θεματολογία. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες και κρατικές αγορές. Α, πώς να το κάνω. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να σας απαντήσω γραπτώς τα ερωτήματά σας, αν επιτρέπετε, να το κάνουμε. Μπορεί έτσι να απαντηθούν τα όσα δεν κατάφερα να καλύψω. Σας ευχαριστώ. We, will come back. Θα επανέλθουμε με γραπτό τρόπο, με γραπτές απαντήσεις σε αυτά. Εντάξει. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα. Να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που ήδη μας έδωσαν κάποιο χρόνο παραπάνω. Ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε, που απαντήσατε στις περισσότερες ερωτήσεις και μας δώσατε την ατζέντα σας, τις ιδέες σας και πολλές απαντήσεις. Εμείς θαυμάζουμε τον ενθουσιασμό σας και τη φιλοδοξία σας και θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να τα επιτύχετε όλα αυτά και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή και θα σας ξανακαλέσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Πριν κλείσουμε τη συνεδρία, να θυμίσω ότι έχουμε μια ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στις 4.30 ε, γιατί θα έχουμε εδώ το πρόεδρο, την πρόεδρο κυρία Τένεμπραουμ τη της Επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου για τα θέματα προστασίας, ε, μάλλον ε, ασφάλειας των προϊόντων των καταναλωτικών. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ.